Hello. Shall we start? Yes, um, you have enough. I think you have enough members. Okay. Um, Mrs. Vice Chair is here. Yeah, anyway, she's there. And I think once you start, then the meeting sort of settles down. Yeah. So, good afternoon, colleagues. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Uh, on item... Θα ξεκινήσουμε αμέσω με το σημείο υπαριθμών 11, κατάρδευση των οδηγιών σχετικά με τη μετρολογία. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Βάις Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι διότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση και αυτό είναι σημαντικό ε, για να μπορέσει ε, το Κοινοβούλιο να καταργήσει έξι οδηγίες για τη μετρολογία και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μία πολύ καλή ε, πρόταση σαν κοινοβούλιο διότι πρόκειται για οδηγίες οι οποίες αναφέρονται σε ε, ε, όργανα μετρήσεως για διάφορες ε, περιπτώσεις όσον αφορά τον βαθμό εινοπνεύματος στα δημητριακά, όσον αφορά διάφορες μετρήσεις τέλος πάντων και θεωρούν ότι αυτές οι οδηγίες μπορούν να καταργηθούν χωρίς να αντικατασταθούν διότι αναφέρονται ε, σε εργαλεία μετρήσεως τα οποία είναι πεπαλαιωμένα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ε, για μία new approach, δηλαδή για μία βελτίωση των τεχνικών ε, προδιαγραφών και απλούστατα θέλω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι διότι θα μπορούσα να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις μου ευθύς εξ αρχής ώστε όταν μας παρουσιάσει το θέμα να περιλάβει και τις απαντήσεις διότι είπατε ότι υπάρχουν τρεις εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες προσφέρονται. Το ένα είναι να παραμείνουμε στο παλιό σύστημα και οι οχτώ οδηγίες να συνεχίσουν να συνεπάρχουν μαζί με ε, τα διεθνή πρότυπα, κάτι το οποίο να πευχόμαστε. Το δεύτερο που πρόκεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διαγραφούν οι οδηγίες αυτές χωρίς να αντικατασταθούν και η τρίτη ε, και εγώ κλείνω υπέρ αυτής είναι ε, να ε, αρθούν ε, δύο-τρεις οδηγίες για τις οποίες όλοι θεωρούμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα είναι όντως πεπαλεωμένος ενώ οι άλλες ναι μεν θα αρθούν αλλά θα ενσωματωθούν στην Measuring Instruments Directives όπου υπάρχει και η νέα προσέγγιση πίεση, πράγμα το οποίο είναι λογικό. Δηλαδή, ε, ε, για να, το να άρουμε τις παλιές ε, προδιαγραφές, συμφωνώ γιατί πρόκειται για παλιά πρότυπα, αλλά θα πρέπει κάπως να ενσωματώνονται ή να συμπεριλαμβάνονται και στο νέο πλαίσιο οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να μας ε, πει ε, ε, για ποιο λόγο καμία εναλλακτική λύση δεν προσφέρει περισσότερες δυνατότητες και παρόλα αυτά η Επιτροπή προτείνει να επιλέξουμε τη δεύτερη εναλλακτική λύση. Ε, επίσης στην προηγούμενη συνεδρίαση ακούσαμε ότι το Συμβούλιο υπάρχει μεγάλη αντιστασή διότι πολλοί είναι κατά της διαγραφής αυτής ε, της ε, κατευθυντήριας γραμμής και της οδηγίας και πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί υπάρχει μία πρακτική εφαρμογή ότι υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές αλλά όχι επαρκής και ε, ή αν μπορούν να μας πούνε ότι αυτό ε, ε, ότι σύμφωνα με την απόφαση του 30, της 30 Σεπτεμβρίου μπορούμε να ξεπεράσουμε τις οδηγίες. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε υψηλότερο επίπεδο προδιαγραφών από ό,τι τα διεθνή πρότυπα και δεν βλέπω λοιπόν πώς αυτό θα επιτευχθεί ε, αν ε, ε, άρουμε τις οδηγίες μας οπότε θα υπάρξει μία καθυστέρηση μέχρι την εφαρμογή των νέων στοιχείων διότι θα ήθελα να ξέρω οδηγία που υπάρχει ένα πρότυπο αν είναι ε, ευρωπαϊκή προδιαγραφή αν προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας νομίζω ότι αυτό το έγγραφο είναι πολύ βασικό και θα χρειαζόμαστε αυτό το έγγραφο για να αποφασίσουμε και να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση όπου θα επιλεχθεί να αρθούν δύο, τρεις και τα υπόλοιπα να περιληφθούν στην οδηγία και να αρθούν μόνο όταν δεν θα δημιουργείται ένα ε, κενό δικαίου και να υπάρξει μια διαθεσμική συμφωνία η οποία θα προβλέπει ότι είναι υποχρεωτική σημαντικό να μην υπάρξει νομικό κενό. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκονται τα κενά, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι 30 Σεπτεμβρίου τέλειωσε η προθεσμία, τι λέγεται στα κράτη-μέλη, ε, διότι ξέρω ότι για ορισμένες οδηγίες λέγουν ότι μπορούν να αρθούν, οπότε θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει η συνεργασία, αλλά θα μας ενδιαφέρει επίσης να μπορέσουμε να βρούμε μία διέξοδο από το τωρινό πρόβλημα και ε, περιμένω με ενδιαφέρον να σας ακούσω. Ευχαριστώ κυρία Βάις Γκέρμπερ. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ε, ο κ. Βινσέντε Λόις Αργουέλε. Euh, Καλημέρα σας. Άκουσα με προσοχή την παρουσίαση της ε, εισηγήτριας. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στη συνεννόηση, αλλά καλό θα ήταν ο Ντανιέλ σε λίγο να μας δώσει περισσότερες ε, λεπτομέρειες, μια και το ζητήσατε και εσείς κυρία εισηγήτρια. Να σας πω κάποια εισαγωγικά στοιχεία πριν παρουσιάσω την μελέτη επιπτώσεων. Πρόκειται για οκτώ οδηγίες για τους μετρητές. Αυτές οι οδηγίες είναι οδηγίες σχεδόν άκυρε σήμερα, ε, χρησιμοποιούνται ελάχιστα σήμερα, γιατί οι τεχνικές μέτρησης έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που αυτό που προβλέπεται σε αυτές τις οδηγίες δεν εφαρμόζεται εκ των πραγμάτων. Παρά τα αυτά, εδώ και κάποια χρόνια δεν υπάρχουν ε, φραγμοί στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Το εμπόριο αυτών των προϊόντων δεν ε, συναντά καμία δυσκολία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Έχουμε τα αποτελέσματα της ε, μελέτης επιπτώσεων, τα οποία δεν μας ε, δεν κινούνται προς τη μία κατεύθυνση ούτε προς την άλλη. Δηλαδή δεν υπάρχει φραγμό στην ελεύθερη κυκλοφορία και πάλι με βάση αυτή τη μελέτη δεν υπάρχει κάποιο διοικητικό πρόβλημα που να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Η Κομισιόν, μια και δεν υπάρχουν καθαρά συμπεράσματα της μελέτης επιπτώσεων, ε, ακολούθησε την αρχή του εφνομοθετήν, της απλούστευσης. Δηλαδή, δεν νομοθετούμε εκεί που δεν υπάρχει λόγος να νομοθετήσουμε. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Γιατί, πώς θα λειτουργούσε η αμοιβαία αναγνώριση αν δεν υπήρχε ε, νομοθεσία εναρμόνισης. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ερώτημα, το θέσατε κι εσείς κύριε Σιγήτρη. Ε, Δυστυχώ ε, την περασμένη φορά δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά νομίζω ότι ακούστηκε. Στην πράξη, σε όλου του τομεί αυτή τη οδηγία έχουμε ήδη διεθνεί κανόνε, διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται και από τα κράτη-μέλη. Εξάλλου είναι υποχρεωτικοί αυτοί οι κανόνε, αυτά τα πρότυπα και που λειτουργούν εξαίρετα. Για να λειτουργήσει καλά η αμοιβαία αναγνώριση, συμφωνώ και εγώ ότι χρειάζεται μία ε, νομοθεσία. Πρόκειται για μετρητές, δεν πρόκειται για οδηγίες που προσπαθούν να εναρμονίσουν συνθήκες ασφαλείας. Προσπαθούμε να εναρμονίσουμε εργαλεία μέτρησης, μετρητές, ούτω ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στις συναλλαγές. Άπαξ και υπάρχει ένας διεθνής κανόνας ε, ή μια, ένας κοινοτικός κανόνας, το άρθρο 28 της συνθήκης ισχύει. Γιατί οποιοδήποτε κράτος μέλος που παίρνει μια νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να την κοινοποιήσει και αν παρελπίδα ε, απόκλινε από αυτή την αναφορά, ούτως ώστε να δημιουργεί φραγμούς, θα έπρεπε να δικαιολογήσει αυτή την απόκληση. Δεν έχουμε παραδείγματα. Παρ' όλα αυτά, καταλήγουμε στο ότι εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη να νομοθετήσουμε πέρα από τους ε, διεθνείς κανόνες, δεν το κάνουμε. Έχουμε τους διεθνείς κανόνες, τα διεθνή πρότυπα, δεν πάμε παραπέρα. Υπάρχει ένας τομέας για τον οποίο δεν υπάρχουν ε, διεθνείς κανόνες. Και είναι ο πιο σημαντικός τομέας ίσως επί του οποίου τα κράτη-μέλη ζητούν μία νομοθεσία στην πλειοψηφία τους. Ε, μιλάμε για τα, για τα μανόμετρα, για τα ελαστικά. Τους μετρητές δηλαδή μέτρησης πίεσης για τα ελαστικά. Δεν υπάρχει σήμερα μια, ένας διεθνής κανόνας που να ικανοποιεί ε, τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν ετοιμάζει μια εντολή για την Επιτροπή α, Ρύθμισης ούτω ώστε να έχουμε αυτή την τεχνική αναφορά που θα ήταν μια κατευθυντήρια γραμμή στο βαθμό που υπάρξει ανάγκη για νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Κάτι που δεν το πιστεύουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν από κοινού με, και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του εφνομοθετή Μα οδηγούν στο να καταλήξουμε ότι σε αυτό το τομέα δεν χρειάζεται να νομοθετήσουμε. Ούτε καν με ένα παράτημα σε μια, για μια μελλοντική α, τροποποίηση. Πιστεύουμε ότι δεν είναι απαραίτητο, αλλά έστω αν χρειαστεί θα ήταν ο πιο ήπιος τρόπος για να το κάνουμε. Μέσω ενός παρατήματος δηλαδή. Αλλά ο ευρωπαϊκός κανόνας που θα αναπτυχθεί με βάση την εντολή της ε, Κομισιόν αρκεί για να εξασφαλιστεί η πλήρης αμοιβαία αναγνώριση. Πολύ ωραία. Θα σταματήσω εδώ. Και αν ε, μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, ο συνάδελφος ο Ντάνιελ θα σας κάνει μια παρουσίαση πιο λεπτομερή. Ο κύριος Χάνικε, ο Ντανιέλ Χάνικε. Thank you. Ευχαριστώ. Έβαλα κάποιες ε, πληροφορίες ε, στις διαφάνειες που προέρχονται από το έγγραφο που υπάρχει και στη διάθεσή σας ε, στην είσοδο του, της αίθουσας και ονομάζεται μελέτη αντικτύπου. Ε, να δούμε ε, τις επιλογές, τις ε, εναλλακτικές λύσεις, τα θέματα τομέα και τα συμπεράσματα. Και στο τέλος θα επανέλθω σε κάποιες ε, ερωτήσεις. Λοιπόν, καταρχάς, ο κύκλος εργασιών. Έξι τομείς είναι. Είναι μικρός ο κύκλος εργασιών. Στα δεξιά σας βλέπετε τη στήλη που φτάνει αθρηστικά στα 40 εκατομμύρια. Ε, αυτά καλύπτουν οι οδηγίες παλιάς προσέγγισης. Η επόμενη στήλη μιλάει για 80 εκατομμύρια εκτός της οδηγίας, έτσι, εκπίπτουν του α, πεδίου εφαρμογή. Τα περισσότερα μανόμετρα ελαστικών εκφεύγουν των οδηγιών αυτή τη στιγμή. Το σύνολο είναι 120 εκατομμύρια. Έχουμε υπό τις οδηγίες 40 εκατομμύρια και εκτός των οδηγιών πιο τεχνικά προηγμένα 80 εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια είναι το σύνολο. Και υπό τις οδηγίες το μεγαλύτερο νούμερο κάτω από τα 40 εκατομμύρια είναι τα 30 εκατομμύρια για τα σταθμά. Ε, για να ζυγίζουμε φορτηγά και τα λοιπά, όχι για τους καταναλωτές, έτσι δεν είναι σταθμά για τους καταναλωτές. Μιλάμε λοιπόν για μικρούς τομείς. Μιλούσαμε, όταν μιλάμε για τις ε, οδηγίες ε, για τους μετρητές, ε, σκεφτόμαστε αρχικά δισεκατομμύρια. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εκατομμύρια. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση σήμερα ουσιαστικά σας την έχω εξήγηση. 40 εκατομμύρια με βάση το, το σήμα συμβατότητα ΕΚ και τα υπόλοιπα 80 εκατομμύρια καλύπτονται υπό την αμοιβαία αναγνώριση. Η αμοιβαία αναγνώριση λοιπόν λειτουργεί στον τομέα, ε, τα κράτη-μέλη νομοθετούν, ρυθμίζουν. Και η τρίτη δυνατότητα είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Και αυτή είναι μια εκτεταμένη κατάσταση, δηλαδή όλα τα προϊόντα ε, είναι δεκτά στην αγορά. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Η επόμενη επιλογή λοιπόν ποια θα ήταν. Θα ξεφορδωθούμε την νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι κρατάω την ίδια σειρά 1, 2, 3. Τι θα γίνει αν ξεφορτωθούμε την παλιά προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να έχουμε εθνικούς κανόνες που να βασίζονται στα διεθνή πρότυπα. Είναι πρότυπα τα οποία ε, ισοδυναμούμε τις οδηγίε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν για όλου του τομεί και επομένω τεχνικώ πώ τίποτα δεν αλλάζει. Το μόνο που θα αλλάξει είναι το σήμα. Ε, ούτως ώστε να αναγνωρίζεται και από τι άλλε χώρε υπό την αμοιβαία αναγνώριση. Η άλλη επιλογή είναι να μην υπάρχουν εθνικοί, εθνικοί κανόνες, πολύ πιθανό και αυτό, γιατί πολλέ από τι οδηγίε και τα μέτρα αυτά ε, είναι απειρχιωμένα. Επομένω, πολλά κρατημέλη μπορούν να ξεφορθούν τα πάντα σε ό,τι αφορά το άλλο κομμάτι που δεν ρυθμιζόταν μέχρι τούδε, δηλαδή των 80 εκατομμυρίων, συγγνώμη, τίποτα δεν αλλάζει. Έβαλε εδώ όλα τα στοιχεία, ούτω ώστε να μπορείτε να καταλάβετε τι γράφει το κείμενο έτσι με απλό τρόπο. Αν πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε την κατάσταση αν ε, νομοθετήσουμε υπό το MID, θα αλλάξουμε τις οδηγίες της παλιάς προσέγγισης και θα τις βάλουμε υπό το Measuring Instrument ε, Directive. Εκεί όμως υπάρχει ένα opt-out. Ε, όσα κρατημέλη λοιπόν δεν θέλουν νομοθεσία, λένε ότι εγώ δεν εντάσσουμε εδώ. Επομένως δεν θα μεταφερθούν στην MID και τα 40 εκατομμύρια. Το κομμάτι που καλύπτεται τώρα από τους ε, εθνικούς κανόνες, εδώ θα έχουμε τις αλλαγές. Ε, αν αφήγουν οι εθνικοί κανόνες ε, και αντικατασταθούν από κανόνες MID. Εδώ μπορούμε να έχουμε ε, σοβαρές αλλαγές για τα κράτη-μέλη που νομοθετούν. Αν δεν υπάρχουν εθνικοί κανόνες, ή μάλλον, συγγνώμη, μπορούμε να πούμε ότι εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο, θα κάνω χρήση του opt-out. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε αυτήν την περίπτωση. Και η άλλη δυνατότητα, εάν δεν έχεις αυτή τη στιγμή κανόνες, Μπορεί να θες να τους έχεις στο μέλλον. Πάλι opt-out. Επομένως, το opt-out είναι μια σοβα... ένα σοβαρό ενδεχόμενο, εάν επανανομοθετήσουμε. Μιλάμε για 120 εκατομμύρια και μόνο ένα μικρό τμήμα ενδεχομένω αυτών των 120 εκατομμυρίων μπορεί να καλυφθεί από μια επανανομοθέτηση. Ε, βλέπετε την τελευταία περίπτωση καθόλου κανόνες. Ε, μπορούμε, να πούμε, μπορούμε να πούμε θα κάνω κανόνες και μπορούμε να πούμε θα χρησιμοποιήσω το opt-out. Αυτά είναι τα διάφορα σενάρια και πάμε τώρα στις επιπτώσεις. Αν κάποιος νομοθετήσει, μπορεί να έχει ε, υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Δεν μιλάμε για ασφάλεια, δεν μιλάμε για τους καταναλωτές. Σχεδόν δεν υπάρχει καμία επαφή με τους καταναλωτές, έτσι. Οι καταναλωτές ε, δεν τα παίρνουν μυρωδιά αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για βιομηχανικούς τομείς, εκτός για τα μανόμετρα ελαστικών, όπου υπάρχει μια επαφή, ας πούμε, όταν πας στο βενζινάδικο και φουσκώνεις τα ελαστικά σου. Επομένως, αν, έχεις, αν έχουμε κανόνες, εθνικούς κανόνες ή οδηγίες, έχουμε υψηλή προστασία, αλλά φυσικά υπάρχει κόστος ε, για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και την εποπτεία της αγοράς. Κάποιος πρέπει να πληρώσει βέβαια, αλλά κάποιος υποφελείται. Επομένως, αθρηστικά φτάνουμε στο μηδέν. Βασικά αυτά βλέπετε σε αυτές τις στήλε. Βλέπετε στην πραγματικότητα ότι αν τις κοιτάξετε ένα δύο, στην αρχή έχουμε το κόστος της νομοθεσίας, εν συνεχεία στη δεύτερη στήλη έχουμε το κόστος της μη νομοθεσίας. Δεν υπάρχει κόστος δηλαδή. Εν συνεχεία, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να κάνουν μάλλον αυτό που κάνουν. Εάν έχουν ρυθμίσεις, θα συνεχίσουν να έχουν. Και αν όχι, δεν έχουν δηλαδή νομοθεσία, θα κάνουν τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση που φαίνεται εδώ. Αν έχεις νομοθεσία πρώτη στήλη και την κρατήσεις που και βασίζεται στα διεθνή πρότυπα, δεν θα έχεις ουσιαστικά καμία αλλαγή στην ε, κατάστασή σου. Σε όλα τα σενάρια μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά αν έχεις νομοθεσία και θες να την κρατήσεις, δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές. Εάν ε, δεν είχες ε, και πάλι opt-out, δεν έχεις κόστος. Τώρα, η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή. Τα κράτη-μέλη θα περάσουν από τη μη νομοθεσία στην νομοθεσία. Ή θα περάσουν από την νομοθεσία στην μη νομοθεσία. Εδώ έχουμε επιπτώσεις. Αλλά είναι μάλλον απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί να αρχίσουν να ρυθμίζουν τώρα πράγματα που δεν είχαν ρυθμίσει ποτέ. Γιατί θα αρχίσουν ξαφνικά να μην ρυθμίζουν τα οποία ρύθμιζαν μέχρι τούδε. Εδώ έχουμε όλες τις ε, πιθανότητες. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε, είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα. Πάμε στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια. Πάμε στα τομεακά θέματα τώρα. Και αυτά είναι ενδιαφέροντα γιατί μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα κάποια μη προφανή πράγματα στα κάθαρτα ύδατα υπάρχει ένα πρότυπο που δεν αναφέρεται στην μελέτη επιπτώσεων. Για, υπάρχει ένα πρότυπο για τα καθαρά ύδατα. Και οι μετρητές ακάθαρτων νερών αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο. Δηλαδή αυτό που έχουμε για τα καθαρά ύδατα ε, υπό το MID, ουσιαστικά το χρησιμοποιούσαμε και για τα κάθαρτα ύδατα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αυτό το πρότυπο για να νομοθετήσουμε σε εθνικό επίπεδο. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για λύματα σε ε, που σε ορισμένε χώρες είναι πολύ σημαντικό και σε άλλες όχι. Ε, παρεκκλήσεις. Ε, χώρες έχουν, ορισμένε χώρες δεν το θεωρούν καθόλου ε, σωστό. Ε, και είναι μικρό και ο κύκλος εργασιών. Επίσης, ε, αποκλείεται να το χρησιμοποιήσουμε στους μετρητές ακάθαρτων υδάτων για τα νοικοκυριά. Τώρα, ε, στην ε, γεωργία χρησιμοποιούμε το πρότυπο ISO. Και χρησιμοποιείται και στους αλκοολομετρικούς πίνακες. Υπάρχει ένα πρότυπο ISO και υπάρχει και στην νομοθεσία την αγροτική. Επίσης, ε, επομένως υπάρχει νομοθεσία για τους αλκοολομετρικούς κανόνες. Αλκοόλ σημαίνει α, όχι μπύρα, σημαίνει α, αλκοολούχα και κρασί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σταθμά. Υπάρχει ένα πρότυπο OML, δεν υπάρχει καμία τίποτα τόμο. 1 ε, κιλό, 10 κιλά, 50 κιλά. Ε, ο κύκλος εργασιών είναι ουσιαστικός, αλλά σε ό,τι αφορά την επαφή με τους καταναλωτές, στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούνται για τους καταναλωτές αυτά τα σταθμά. Ουσιαστικά ε, ζυγίζεται τα, τα τρόφιμά σας, ας πούμε, σε μία αυτόματο, αυτόματη ζυγαριά. Εν συνεχεία, πάμε στους μετρητές ε, πίεσης ελαστικών. Ε, αυτό είναι σημαντικό, το IML. Ε, θα υπάρξει πολύ μεγάλη τεχνική πρόοδος, γιατί στο 2014 όταν νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή θα έχουν ένα σύστημα διαχείρισης της μέτρησης των ελαστικών. Και για κάθε ελάστιχο θα έχουμε μία ένδειξη εάν η πίεση του ελαστικού είναι σωστή ή όχι. Φυσικά υπάρχουν διάφορα TPMS. Γι' αυτό υπάρχει και παγκόσμιο πρό, ε, πρότυπο για τα TPMS. Γι' αυτό ε, θέλουμε να εκδώσουμε μια εντολή ε, για, τα πρότυπο, για ένα πρότυπο και θέλουμε το εξή. Αν παραδείγματο χάρη τα λάστιχά σα δεν είναι καλά, ε, και χτυπάνε, χτυπάει ένα καμπανάκι ας πούμε, στο αυτοκίνητο συνέχεια επειδή η πίεση των ελαστικών δεν είναι καλή, αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τομεί, ε, αναπτύσσεται και δεν ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει. Ε, έχει νόημα να αρχίσουμε να νομοθετούμε, διερωτόμαστε τώρα το, η Κομισιόν, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ υπάρχουν τεχνικές λύσεις που αλλάζουν, συζητιώνται, ε, τα πράγματα κινούνται. Και όταν εμείς τελειώσουμε, ίσως ε, κάθε αυτοκίνητο που θα παράγεται θα έχει ένα TPMS. Επομένως, νομίζουμε ότι καλό θα ήταν να έχουμε ένα πρότυπο ισότιμο και οποιοδήποτε θέλει να νομοθετήσει να ακολουθήσει αυτό το πρότυπο. Τώρα, αν αποδειχθεί ότι θα χρειαστούμε νομοθεσία για κάποιο λόγο, τότε φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε ανοιχτοί. Τίποτα δεν αποκλείεται στα MID μπορούμε να προσθέσουμε νέα παραρτήματα σε αυτές τις οδηγίες για τους μετρητές. Μετά, η, μάζα των σιτηρών. Έχουμε ένα πρότυπο OIML, αλλά η νομοθεσία για τα γεωργικά αναγνωρίζει μόνο το πρότυπο ISO. Είναι πολύ σημαντικές μετρήσεις αυτές για τους γεωργούς, για να πληρωθούν τα χρήματα. Επομένως, ε, αυτό που έχει σημασία για μας είναι ο μικρό κύκλο εργασιών. Και ένα πολύ δύσκολο θέμα. Αν το ρυθμίσουμε, αν υπάρξει νομοθεσία υπό το MID, τι θα κάνουμε την γεωργική νομοθεσία. Θα πρέπει να στείλουμε ένα email και να πούμε εμείς έχουμε νομοθεσία, προσαρμόστε την νομοθεσία σας. Επομένως, είναι δύσκολο να αρχίσουμε τώρα να νομοθετούμε. Ε, το ίδιο πρόβλημα το έχουμε και, στο, και στα αλκοόλ. Έπειτα, για τις δεξαμενές ε, πλοίων υπάρχει ένα ε, πρότυπο OIML, δεν υπάρχει καινοτομία. Αυτά τα, αυτές οι δεξαμενές ούτως ή άλλως δεν χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές, ε, γιατί κανείς δεν τις εμπιστεύεται. Παραδείγματος χάρη αντλείς, βάζεις πετρέλαιο σε ένα πλοίο, το, πλοίο χρησιμοποιείται, το χρησιμοποιεί αυτό το πετρέλαιο και μετά το βγάζουμε. Πώς το τσεκάρουμε. Όταν μπαίνει το, το πετρέλαιο στην δεξαμενή, το μετράμε και συνεχεία όταν βγάζουμε το πετρέλαιο μετά το τέλος της, του ταξιδιού ας πούμε, ε, βλέπουμε πόσο, βλέπουμε αν κάνουμε την αφαίρεση, πόσο έχει καταναλώσει το πλοίο. Δεν θεωρούμε λοιπόν ε, ότι θα πρέπει αυτά, αυτές οι δεξαμενές να είναι αντικείμενο τυποποίησης. Είναι ένα από τα πολλά στοιχεία σε ένα πλοίο. Και η οδηγία για την ασφάλεια στη θάλασσα δεν θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τα υπάρχουν θα υπάρχουν τα πρότυπα που έχουμε στον κανονισμό. Και επιπλέον είναι και μικρός ο κύκλος εργασιών. Λειτουργούμε με ευρωπαϊκά πρότυπα που είναι θελοντικά. Όποιο θέλει να τα χρησιμοποιήσει, τα χρησιμοποιεί. Τώρα στο έγγραφο με τα βασικά θέματα σας δίνουμε μια επισκόπηση ε, με τις απόψεις των κρατών μελών. Το είχατε ήδη αυτό από το Μάιο του 2008. Αυτός ο πίνακας ε, μοιάζει πολύ με τον επικυροποιημένο ε, που επικυροποιήθηκε ε, συγγνώμη, το Φεβρουάριο του 2009, πίσω από την πλάτη της Προέδρου. Αυτή είναι η κατάσταση στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου, η τρέχουσα κατάσταση. Η σιωπήρη πλειοψηφία στο Συμβούλιο είναι υπέρ της ανάκλησης των περισσότερων οδηγιών ακόμα. Παντού βλέπετε υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ της ανάκλησης εκτός από τα μανόμετρα ελαστικών. Στο σημείο 6 δηλαδή. Έχετε μια πλειοψηφία 15 κρατών, εκεί, για τα μανόμετρα. Από την άλλη, Α, τότε βέβαια δεν ξέραν ότι ε, δουλεύαμε για μία εντολή για τα μανόμετρα. Μπορεί να υπάρξει αλλαγή λοιπόν, θα πρέπει να το τσεκάρουμε. Επίση υπάρχει μια μειοψηφία μπλοκαρίσματο σχεδόν παντού. Μια μειοψηφία άρνηση ε, κυρία. Δεν φαίνεται από αυτά τα νούμερα, αλλά το επιβεβαιώνω ότι υπάρχουν σχεδόν παντού τέτοιου τύπου ε, μειοψηφίε. Ποιο είναι ο γενικό, το γενικό πλαίσιο. ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα για τις οδηγίες, πρέπει να μπείτε στις λεπτομέρειες. Εδώ θα επισέλθω και στις ερωτήσεις ε, της εισηγήτριας. Δουλεύει αμοιβή αναγνώριση. Εδώ βάλαμε κάποιες προϋποθέσεις που είναι σημαντικές για την ε, αμοιβή αναγνώριση προκειμένου να είναι λειτουργική. Φυσικά αυτό ε, συνδέεται με την ε, επικουρικότητα, με τις εθνικές επιλογές. Α, επιλέγεις, θες να έχεις νομοθεσία ή δεν θέλεις. Περιοδικός έλεγχος. Είναι πολύ σημαντικός με αυτά τα μέσα. Είναι πάντα εθνικοί κανόνες. Δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι περιοδικοί έλεγχοι. Ούτε στην οδηγία για τους μετρητές, ούτε στην άλλη οδηγία. Υπάρχει μια εθνική προτίμηση για ρύθμιση ή όχι, ή για περιοδικούς ελέγχου ή όχι. Ε, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, εθνικής επιλογής, παράδοση αλλά και επιλογής. Αν κάποιο πει ότι ε, είναι επικίνδυνο να μην ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών τακτικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να στείλει δηλαδή ένα κράτο μέλο έναν εμπειρογνώμα στι Βρυξέλλε για να ζητήσει κάτι τέτοιο περιμένουν ε, στη χώρα τους και δεν θα ζητήσουν, δεν θα έρθουν στις Βρυξέλλες εδώ για να ζητήσουν το κάνουν, θα κάνουν κάτι στη χώρα τους. Τα διεθνή πρότυπα επίσης πρέπει να υπάρχουν για να βασίζουμε τους κανόνες μας και τους νόμους μας πάνω. Ε, είναι αυτά που απαιτεί ο ε, ΠΟΕ και τα TBT. Θα με εξέπλητε ε, αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτό που θέλει μια χώρα και των διεθνών προτύπων. Ε, μάλλον ξέρω μία διαφορά. Ε, γλωσσικές απαιτήσει. Υπό το MID έχουμε πολύ αυστηρές απαιτήσει ε, για τη γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 32 διαφορετικά πρότυπα για τις γλωσσικές απαιτήσει. Ε, μπορεί κάθε χώρα να απαιτήσει η γλώσσα της να είναι πάνω στις οδηγίες. Επομένως, ε, υπό το MID Ε, έχουμε κάτι το οποίο συμφωνεί απόλυτα με τον ΠΟΕ και το TBT. Τίποτα δεν θα ήταν περίεργο ε, με το να έχουμε εθνικές ας πούμε οδηγίες, μάλλον να έχουμε οδηγίες ε, στην εθνική γλώσσα, στην εθνική γλώσσα τα μανόμετρα. Το βάλαμε λοιπόν στο MID και κανένας δεν έφερε αντιρρήσεις στον ΠΟΕ. Και ούτε εμεί δημιουργούμε προβλήματα σε άλλε χώρε που θέλουν να βάλουν ε, τη γλώσσα του. Να ένα καλό παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει ένα κράτο μέλο αν θέλει να προχωρήσει σε εθνικού κανόνε. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια βέβαια στο εμπόριο και αυτό βασίζεται και στη συνθήκη. Επομένω θα πρέπει να γράψει του νόμου σου και να λε ότι δεχόμαστε ε, τα προϊόντα που γίνονται αλλού εάν είναι εξίσου, έχουν εξίσου καλέ ε, επιδόσει. Αυτά βασίζονται ε, στα άρθρα 28 έως 30 της συνθήκης. Ε, υπάρχουν χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων νομολογίες, επομένως όλα είναι ξεκάθαρα. Το ίδιο ε, για την αποδοχή της αξιολόγησης συμμόρφωσης. Ε, με πολλούς εθνικούς κανόνες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λειτουργεί. Ε, ένα από τα ενδιαφέροντα πορίσματα ε, της μελέτης επιπτώσεως είναι ότι κανένα δεν μα είπε ότι υπάρχουν εμπόδια στο εμπόριο και ότι δεν υπάρχει αποδοχή τη ε, συμμόρφωση. Αν υπήρχε πρόβλημα θα είχε ε, διαφανεί στη δημόσια διαβούλευση κάπου. Όμως κανένας δεν είπε τίποτα. Ε, και η οργάνωση η Wellmec, που, ε, όπου έχει μια νομοθεσία για συμφωνίες ε, ε, εγκρίσεως τύπου. Εκεί συμμετέχουν όλα τα εθνικά Ινστιτούτα Μετρολογίας κτλ. Και, βασίζονται στα εθνικά, στους, στους διεθνείς κανόνες. Αυτό αναφέρεται στη σελίδα 4 της μελέτης επιπτώσεων. Η Επιτροπή σας πριν από λίγα χρόνια εξέτασε προσεκτικά τον κανονισμό για τη βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ο κανονισμός τώρα ισχύει. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ξεφύγει τους κανόνες της αμοιβαίας αναγνώρισης, οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να ξεφύγει, θα πρέπει εκείνη να αποδείξει ότι έχει δίκιο εναντίον, σε, σε, αντιδιαστολή με τον, με τον ενάγοντα, ας πούμε. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά τώρα για την αμοιβαία αναγνώση, από ήταν πριν λίγα χρόνια. Και τώρα φτάνουμε στα συμπεράσματα τη μελέτη επιπτώσεων. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση που να, προ... να είναι προτιμητέα. Το είπε και η συγγήτρια. Συνήθω ψάχνουμε να δούμε πώς θα νομοθετήσουμε, έτσι. Αλλά όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, Δεν σημαίνει βεβαίως ότι η νομοθεσία είναι κακό πράγμα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχουν ωφέλη, δεν υπάρχουν ε, φραγμοί στο εμπόριο που θα βοηθούνταν να αρθούν ενώ χάρη στην νομοθεσία. Επομένως δεν έχουμε καμία προτίμηση προς την μία προς την άλλη κατεύθυνση. Επιλέξαμε την εναλλακτική λύση 2. Γιατί αυτές οι οδηγίες ούτως ή άλλως είναι απαρχαιωμένες. Ε, πριν από 20 χρόνια ίσως ήταν λιγότερο ξεπερασμένες ε, και 10 χρόνια μετά θα είναι ακόμη περισσότερο Τώρα υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά ε, διεθνή πρότυπα που ισοδυναμούν με τις οδηγίες παλιάς προσέγγισης. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε 27 διαφορετικά καθεστώτα. Ούτω ή άλλω τα διεθνή πρότυπα είναι εξίσου αυστηρά με τι ε, οδηγίε ε, παλιά προσέγγιση. Επομένω, δεν υπάρχει κανένα λόγο τώρα ξαφνικά τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν διαφορέ. Φυσικά θα μπορούσαν και υπό την ε, παλιά προσέγγιση να έχουν εναλλακτική νομοθεσία και κάποιοι έχουν πιο αναπτυγμένη νομοθεσία, πιο αναπτυγμένα εργαλεία και μέσα. Αλλά ακόμα και έτσι δεν, έχουμε, δεν μας έχουν αναφέρει πουθενά ε, φραγμό στο εμπόριο. Επομένως μπορεί να έχεις εθνικούς κανόνες, να αναγνωρίσει τα πρότυπα παίζω για τα αλκοολόμετρα, ας πούμε. Αλλά κανένα δεν μα είπε ότι δημιουργήθηκαν φράγμοι στο εμπόριο σε αυτήν την περίπτωση. Επομένω, δουλεύει αν δεν αναγνώρισε από ό,τι φαίνεται. Είναι μικρή τομή σε σχέση με άλλου στον, στον MID. Δεν υπάρχει μεγάλη επαφή με του καταναλωτέ. Α, προσπαθώ να διαβάσω και την τελευταία πρόταση που δεν τη βλέπω όμως. Α, το opting out. Μπορούμε να το περιμένουμε αυτό. Σας είπα τα αριθμητικά στοιχεία στους προηγούμενους πίνακες για τα κράτη-μέλη. Το opt-out πρέπει να το περιμένουμε. Δεν υπάρχει μεγάλη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών ότι αυτή είναι η νομοθεσία που χρειάζονται για τους τομείς αυτούς. Νομίζω ότι αρκούν αυτά, θα ακούσω σχόλια τώρα και μπορούμε να επανέλθουμε. Να επανέλθω εγώ δηλαδή, αν μου κάνετε ερωτήσεις. Many thanks for this profound... Ευχαριστώ πολύ για αυτή την διεξοδικότατη επεξήγηση. Βέβαια είμαι βέβαιη ότι τα, της μετρολογίας δεν τα καταλαβαίναμε πριν, τώρα είναι σαφή. Έχω αρκετούς ομιλητές. Πρώτη, κυρία Γκέρχα. Ευχαριστώ. Όντως ήταν τόσο σαφές, ώστε είχα δυσκολία να παρακολουθήσω, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, δεν παρακολουθώ την λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορώ να παρακολουθήσω διότι εδώ λέγεται ότι υπάρχουν εναρμονισμένες οδηγίες, δεν υπάρχουν εμπόδια στην αγορά για το εμπόριο, ως εκ τούτου πρέπει να διαγράψουμε αυτούς τους κοινούς κανόνες. Είναι μια λογική η οποία μου διαφεύγει διότι σε πολλές περιπτώσεις όντως υπάρχουν πεπαλαιωμένες ρυθμίσεις και αυτό το δέχομαι. Αυτό το οποίο με ενοχλεί όμως είναι με τον κατάλογο τον οποίο επιτέλους έχουμε για να δούμε τι καθεστώς ισχύει στις διάφορες χώρες να βλέπουμε ότι εκτός μίας περίπτωσης υπάρχει μία, ε, ε, μία μειοψηφία κατά αυτής της, ε, αυτής της διαγραφής. Οπότε υπάρχει μόνο μία περίπτωση και ελπίζω ότι στο ερώτημα θα απαντήσει το Συμβούλιο ποιοι είναι οι λόγοι. Διότι αν είναι τόσο πεπαλαιωμένες αυτές οι ρυθμίσεις και τόσο πια ε, ξεπερασμένες και δεν παίζουν κανένα ρόλο στην ε, βιομηχανία μας, τότε δεν πρέπει να υπάρχει και αντίρρηση. Και αυτό δεν το βλέπω. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν τόσα κράτη τα οποία είναι κατά της διαγραφής. Το δεύτερο θέμα, το οποίο επίσης μου διαφεύγει, είναι ότι είπατε κάτι, ότι δηλαδή όπου θα μπορούσε να υπάρξουν κενά για τις κυβερνήσεις μπορεί να ισχύσει το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης. Το πρόβλημα με την αμοιβαία αναγνώριση είναι ότι αυτή βασίζεται στο εθνικό δίκαιο. Δηλαδή, ουσιαστικά αντικαθιστούμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό ενδεχομένως με 27 νομοθετήματα αν υπάρχει κάποιο κενό. Αναρωτιέμαι, είναι ο σωστός τρόπος λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της εισηγήτριας, δηλαδή να κοιτάξουμε κάθε οδηγία διεξοδικά, να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε οδηγία που και μέσω ποιων κανόνων ISO του ΠΟΕ ή άλλων καλύπτεται και μπορεί πλέον να διαγραφεί. Και επίσης είπατε ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τη σήμανση διότι όταν μιλάμε για σήμανση είναι ακριβώς ε, μία από τις βάσεις ε, συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει ενιαία σήμανση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί προτού διαγράψουμε τις ε, οδηγίες, γι' αυτό και εγώ λέω ότι το δεύτερο θέμα που ανέφερε η κυρία Βάις δηλαδή ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να τις, ε, μετα, ε, ε, να ενσωματώσουμε στην ρύθμιση την ενιαία η οποία θα γίνει πως αυτός δεν θα ήταν ο καλύτερος τρόπος και ο πιο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Με ενοχλεί κάπως διότι είπατε παρόλο που το βρήκα συμπαθητικό ότι όσον αφορά τα όργανα μετρήσεως των ελαστικών μέχρι το 2014 θα έχουμε αυτό το ενιαίο νέο σύστημα και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά με συγχωρείτε, 2014 μου λέτε δηλαδή ότι ως τότε έχουμε μπόλικο καιρό. Δηλαδή θα έχουμε τα ενιαία τα νέα, ε, νέους τρόμπς μετρήσεως αλλά δεν θα έχουν εξαφανιστεί όλα τα παλιά αυτοκίνητα. Η μαμά μου έχει ένα αυτοκίνητο 11 ετών και θα συνεχίσει να το έχει όσο ζει. Οπότε υπάρχει ακόμη ένα μεσοδιάστημα. Τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα αυτό όπου θα υπάρχουν τα παλιά, ε, ε, τα παλιά αντικείμενα. Οπότε εγώ θα έλεγα να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο οποίον πρότεινε η συγγήτρια. Δηλαδή, να κοιτάξουμε μία-μία τις οδηγίες να δούμε αν υπάρχει νόημα να τις διαγράψουμε και να τις καταργήσουμε οπότε θα το πράξουμε ή ε, αν πρέπει να ενσωματωθούν στην ενιαία οδηγία τότε αυτό να το πράξουμε ακόμη ε, και αν ε, όταν υπάρχουν επουσιώδεις ε, δεν είναι κριτήριο για μένα αυτό ή θα αποφασίσουμε να την αναμορφώσουμε ή να την διατηρήσουμε και αυτές είναι οι αλλαγές τις οποίες προτείνω. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι είναι ενθουσιασμένοι και παθιασμένοι με την μετρολογία. Τώρα ο κύριος Μπουρζουά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι μετά από την παρουσίαση η κατάσταση δεν είναι πιο σαφής για μένα και όχι γιατί είχε πολλά ακρόνημα η παρουσίαση, αλλά γιατί η κατάσταση είναι λίγο θολή. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας να μας εξηγήσετε, τουλάχιστον για τις πιο σημαντικές ε, από αυτές τις οδηγίες, γιατί 7 ή 8 ή 10 κράτη-μέλη είναι κατά. Γιατί, γιατί είναι σημαντικό εάν υπάρχουν ε, σοβαροί λόγοι, θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Σε γενικές γραμμές, άποψή μου είναι να ακολουθήσουμε την ε, οδό της απλούστευσης. Αν δεν υπάρχουν φραγμοί για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ε, απλουστεύσουμε την ε, νομοθεσία θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την απλούστευση, τα διεθνή πρότυπα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν πολύ καλά επιχειρήματα προκειμένου να λάβουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Και σήμερα, παρά το γεγονό ότι υπάρχουν κάποια επιχειρήματα, δεν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι αυτή είναι η οδός που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Κυρίως για την ε, πίεση των ελαστικών θα πρέπει να κάνουμε μια πιο διεξοδική συζήτηση. Αυτό είναι σαφές. Όπως είδα και από την παρουσίαση, ε, μιλάμε για ένα τομέα στον οποίο οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σημαντικές. Όχι τεράστιες, αλλά σημαντικές. Και επίσης θα πρέπει να δούμε γιατί κάποια κράτη-μέλη είναι κατά της ανάκλησης κάποιων άλλων οδηγιών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, τότε να τις ε, καταργήσουμε όλες και να πλουστεύσουμε την ε, νομοθεσία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η στιγμή να αποφασίσουμε γιατί δεν έχουμε όλες τις συνιστώσεις. Ευχαριστώ. Ίσως η Επιτροπή μας θα πρέπει να αποφασίσει ε, για ποιο λόγο θεωρούμε ότι είναι διστακτικά κάποια κράτη-μέλη. Είναι γιατί υπάρχει κάποιος εμπειρογνώμενος που απλά θέλει να κρατήσει τη δουλειά του. Για σκεφτείτε το κι αυτό. Ε, να του απολύσουμε τότε. Η κυρία Ρούλα. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι ποιος θα υποφεληθεί από αυτό, γιατί με εκπλήσει ότι κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ζητήσει να γίνει αυτή η απλούστευση. Ποιος το επιθυμεί δηλαδή. Και αν δούμε τη μελέτη των επιπτώσεων δεν βλέπουμε ούτε προτέρημα, ούτε αλλαγή, ούτε τίποτα. Όλα οι απαιτήσει μένουν οι ίδιες. Αλλά ορισμένες χώρες θα το συζητήσουν στο Συμβούλιο και θα έχουν ασχοληθεί με κάτι που κανένα, ε, σε κανέναν δεν ωφελεί, αλλά τελικά θα έχουμε απασχοληθεί με κάτι. Πρέπει να σας πω ότι η ε, απλοποίηση δεν έπρεπε να οδηγεί σε γραφειοκρατική επιβάρυνση. Πρέπει να ξέρουμε γιατί κάνουμε, ό,τι κάνουμε και να αποφασίζουμε. Ο κύριος Κοζούσνιτ. Μπράβο, το, το, είπατε θαυμάσια. Κυρίες και κύριοι, νόμιζα ότι θα τα κατάφερνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν προσφέρεται μια καλύτερη κατάσταση για την μείωση της γραφειοκρατίας παρά όλο να συζητάει κανείς μία ώρα μετά το μεσημεριανό φαγητό με πολλά άδεια έδρανα ένα θέμα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί ε, προς την κατεύθυνση που είπαμε, να αναλύσει κάθε οδηγία χωριστά, να τονίσει και να ερευνήσει ποια είναι η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και μετά να αποφασίσει για να μην προκύπτει το ίδιο θέμα κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. Έχουμε... Κυρία Βάισκερ, θέλετε να μιλήσετε αμέσως, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ. Ε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για τα σχόλια των συναδέλφων και τη στήριξη και έχω να διατυπώσω μία πρόταση. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ ε, εντυπωσιάστηκα με το θέμα της σημάνσεως γιατί το είδα από τα έγγραφα διαφόρων κρατών μελών και είναι ένα θέμα το οποίο ε, ε, πρέπει να κοιτάξω. Γιατί χρειαζόμαστε τη σήμανση των εργαλείων μέτρησης όταν ε, πλέον δεν υπάρχει τίποτα να μετρήσουν. αλλά νομίζω όσον αφορά τα πιεσόματρα για τα ελαστικά είναι κάτι διάζων ήταν το μόνο σημείο επί του οποίου η πλειοψηφία των κρατών μελών ήταν αντίθετη και ε, από εκεί και πέρα ε, ε, οι διάφορες ρυθμίσεις στο γεωργικό τομέα μπορούν να αντικατασταθούν. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι από πλευράς της Επιτροπής, δηλαδή ο πρόεδρος της Επιτροπής ενδεχομένως μαζί μου, να καταρτήσει μία πρόταση και επιστολή στην Σουηδική Προεδρία όπου θα λέει σαφώς ότι ζητάμε να μας πούν για ποια οδηγία και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να παραμείνουν αυτά, αυτές οι οδηγίες διότι ορισμένοι δεν ήθελαν ούτε να το ακούσουν και δεν θα βοηθήσουν. Ε, σήμερα ας πούμε η υπεύθυνο είχε ραντεβού με τον ε, πρέσβη της και δεν μπορούσε να ασχοληθεί αλλά καλό θα ήταν να μας πούν για γιατί σε διαφορετικές οδηγίες επιμένουν ορισμένοι να παραμείνουν οι οδηγίες. Έχει όντως λήξει η προθεσμία, δεν ξέρω τι έχει γίνει εντωμεταξύ, εσείς θα ξέρετε. Ε, παραδείγματος χάρη για την μελέτη επιπτώσεων για το MIB, νομίζω ότι υπάρχει μία αντίσταση, αλλά ακόμη δεν έχω αντιληφθεί γιατί ιδίω ε, γιατί υπάρχει το θέμα αυτό σε κάθε μεμονωμένη ε, οδηγία. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι είχα κατά νου ε, στις 16 Οκτωβρίου να υποβάλω την έκθεσή μου, αλλά νομίζω ότι τώρα έχουμε χρόνο και καλύτερα να το παιδέψουμε λίγο παραπάνω. Να συμφωνήσουμε δηλαδή για ένα ε, διάγραμμα, να κάνουμε μία επιστολή προς τη Σουηδική Προεδρία και να ρωτήσουμε ποια είναι τα αντιεπιχειρήματα σε κάθε οδηγία και να κοιτάξουμε, ε, να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγία προς οδηγία τι συμβαίνει, να ξανασυζητήσουμε το θέμα και μετά εφόσον συμφωνήσουμε βλέπουμε. Ε, ναι μεν ναι, ναι, να καταργηθούν οι παλιές αλλά αυτές οι οποίες χρησιμοποιούνται ακόμη να ισχύσουν. Αυτή είναι μια δυνατότητα κυρία Πρόεδρε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε έτσι και καταρχήν να επέμβουμε στο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή διότι πρέπει να μας δώσουν πληροφορίες τις οποίες χρειάζομαστε ακόμη. Θα ήθελα να ακούσω την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κυρίου Χάνεκ. Πώς αξιολογείται την κατάσταση, ιδίω όταν λέτε ότι ρωτάτε τα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μας περιγράψετε τι σας λένε. Ευχαριστώ. Δύο λόγια θα πω εγώ και θα δώσω μέσα το λόγο στον Τανιέλ. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικό αυτό το ερώτημα. Τα κράτη-μέλη ε, που θέλουν να κρατήσουν αυτή την οδηγία, γιατί τη θέλουν. Ποια είναι τα επιχειρήματα που κρύβονται από πίσω. Θέσαμε το ερώτημα, όχι τώρα, εδώ και καιρό. Και εν συνεχεία θα, ο Ντανιέλ θα σας εξηγήσει τις λεπτομέρειες των απαντήσεων των κρατών μελών. Αλλά πραγματικά δεν θεωρούμε ότι χρήζουν, ότι υπάρχει λόγος για τη χρήση, για, την ασ... για λόγους ασφάλειας, φερρυπίν, για οποιοδήποτε λόγο. Για να διατηρηθούν αυτές οι οδηγίες. Συμφωνώ με όλα τα επιχειρήματά σας. Αλλά η Κομισιόν με όλα αυτά τα δεδομένα ε, καταλήξω συμπέρασμα δεν υπάρχει κανένας λόγος για να προβούμε σε νομοθεσία. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια των βουλευτών και, και, και όλους ιδιαίτερος με κάποια... Έχουμε, 100, έχουμε να κάνουμε 120 εκατομμύρια ευρώ, α, κύκλος, κύκλο εργασιών. Ε, τα 80 εκατομμύρια είναι εκτός των οδηγιών. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από τη μία έχουμε 8 οδηγίες που εφαρμόζονται ελαχιστότατα γιατί οι περισσότερες έχουν συμπληρώσει μια 20 Ο κόσμος ε, έχει αλλάξει άρδιν εδώ και 20 χρόνια. Τι κάνουμε, τις κρατάμε, τις ε, εξυγχρονίζουμε ή τις καταργούμε. Όταν βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη, ε, το συμπέρασμα τη Κομισιόν είναι ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να τι κρατήσουμε. Επομένω, να καταργήσουμε την γραφειοκρατία. Τέλο πάντων, δεν είναι απαραίτητο. Αλλά συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι τα επιχειρήματα των κρατών μελών για να τι διατηρήσουμε. Για τη σήμανση. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ούτω ή άλλω θα υπάρχει μια αναφορά ε, σε κάποιο κανόνα στο προϊόν. θα είναι ε, ε, μια σήμανση που θα παραπέμπει στο πρότυπο και όχι στην οδηγία. Ούτως ή άλλως, ο για τον καταναλωτή που θα είναι ο τελικός καταναλωτής, θα υπάρχει μια αναφορά στη σήμανση. Ούτως ή άλλως, όντως, θα αντικαταστήσουμε μια σήμανση με μια άλλη. Και η ημερομηνία 2014 ισχύει μόνο αν ομοθετήσουμε. Γιατί ο κόσμος, ο τεχνικός, ε, εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από εμά. Νομίζω ότι πολύ πιο γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα να αφήσουμε τους τεχνικούς να δουλέψουν, ε, τους ΕΝ ή οποιοδήποτε άλλου οργανισμού. Επί των λεπτομεριών συμφωνώ, συμφωνώ Κύριε Άρου, λέτε ότι δεν χάνουμε το χρόνο μας, αλλά πραγματικά καλό είναι να δούμε ένα-ένα τα επιχειρήματα και να τα αναλύσουμε. Και μαζί σας και προφανώς με τα κράτη-μέλη. Ο Ντανιέλ θα προσθέσει κάτι. Mr. Ναι, κύριε Hanekak, θέλετε να απαντήσετε σε αυτές τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ευχαριστώ. Κατανοώ πολλά από αυτά που άκουσα εδώ. Σας διαβεβαιώ ότι εργάζομαι 10 χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα, επομένως λίγο πολύ επιρρογνώμονας είμαι, παρόλο που και εγώ δεν καταλαβαίνω πάρα πολλά για το θέμα, αλλά για την οδηγία αυτή ποτέ στα 10 χρόνια δεν άκουσα τέτοια ερώτηση. Είναι η πρώτη φορά που αρχίσαμε ε, να το εξετάζουμε και είπαμε ότι στη φάση της απλούστευσης πρέπει να κάνουμε κάτι, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν 8 οδηγίες και πρέπει να τις καταργήσουμε. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα με του εμπειρογνώμονε, ε, οι πολλοί από αυτού συμμετέχουν και στι ομάδε εργασία του Συμβουλίου, είναι ότι ούτε και αυτοί ήξεραν τίποτα. Οι δεξαμενέ πλοίων, για παράδειγμα, ήταν το απόλυτο κενό. Κανεί δεν ήξερε τι ήταν. Συμφωνώ λοιπόν με πολλά από αυτά που άκουσα εδώ σήμερα. Αν είχαμε πληροφορίε, θα σα τι δίναμε και ποτέ δεν είχαμε πρόθεση να κρύψουμε πράγματα. Στην ε, αξιολόγηση αντικτύπου ε, ακολουθήσαμε τα παραδείγματα που μας έδωσαν οι σύμβουλοι για να εξετάσουμε κάποια παραδείγματα, γιατί δεν υπήρχαν άνθρωποι με εμπειρογνωμοσύνη στο θέμα. Έκτοτε βέβαια κάναμε μια πρώτη καταμέτρηση, είχαμε και τον πύλακα που σας έδειξα, ε, λίγο λιγότερες χώρες, αλλά λίγο πολύ το ίδιο ήταν το τοπίο. είχαμε και ελάχιστα κίνητρα. Κάποια από αυτά τα κίνητρα αναφέρονται στις τελευταίες δύο διαφάνειες. Με χαρά να στα, στα αναφέρω. Ένα που άκουσα έχει να κάνει με τις οδηγίες, γιατί αυτή τη στιγμή λέμε δεν έχουμε φραγμούς ε, στο εμπόριο. Αυτό είναι ένα επιχείρημα. Όντως, αλλά εξακολουθούν να είναι παροχημένα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν φραγμοί στο εμπόριο και στον τομέα στον οποίο δεν υπάρχει ρύθμιση. Ε, στον τομέα στον οποίο υπάρχει τεχνολογία που είναι πολύ πιο προηγμένη. Μιλάμε για ψηφιακά πιεσόμετρα για ελαστικών. Τα βλέπετε στο Βέλγιο παντού και εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Η πρώτη μου αντίδραση λοιπόν ήταν ότι μια χαρά είναι, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία γιατί είναι ψηφιακά, αλλά λειτουργούν μια χαρά. Καλό θα ήταν λοιπόν να ακούσουμε και με κάποιο, από κάποιον που έχει πείρα. Ρωτήσαμε για παράδειγμα άτομα τα οποία έχουν σχετική πείρα με το TPMS. Πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν τα ψηφιακά, ποια είναι η διαφορά τους με τα μη ψηφιακά, τα μηχανικά που περιλαμβάνονται στην οδηγία. Είναι εξίσου ακριβή. Μπορεί και να είναι, αλλά μπορεί και όχι. το γεγονό ότι μπορεί να οδηγήσουν σε νέο φραγμέ στο εμπόριο. Πολύ καλό επιχείρημα, αλλά γιατί. Αν ε, τα διεθνή πρότυπα είναι ήδη με τι οδηγίε, γιατί να οδηγήσουν σε νέου φραγμού στο εμπόριο. Αν δεν υπάρχουν φραγμοί εκτό οδηγίε, γιατί θα έχετε νέου φραγμού μέσω εθνική νομοθεσία. Τα κράτη-μέλη έχουν άδεια να νομοθετούν 30 ε, χρόνια εκ παραλίλου με τις οδηγίες και δεν φαίνεται να δημιουργήθηκαν φραγμοί στο εμπόριο. Υπάρχει ανάγκη να εναρμονίσουμε ε, τεχνολογικώς πιο προηγμένα πρότυπα. Μπορεί, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Το να αρχίσουμε να, να εναρμονίζουμε γιατί αλλάζει τεχνολογία, καταλαβαίνετε πόση δουλειά σημαίνει αυτό για μας. Και για την ανάκλησή τους. Δεν ε, λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες πολιτικές. Ναι, αλλά ποιες είναι οι ανάγκες πολιτικής. Εσείς είπατε ένα-δυο πράγματα εδώ, αλλά είναι όντως ανάγκες πολιτικής. Γιατί δεν τις ακούσαμε σε πιο πρώιμο στάδιο όταν έγινε η δημόσια διαβούλευση. Γιατί δεν ακούσαμε αυτές τις ανάγκες πολιτικής. Υπήρχε για παράδειγμα μία ανάγκη για το περιβάλλον, για, τα, για την πίεση των ελαστικών. Αλλά αυτό καλύπτεται από την οδηγία για την ασφάλεια. Πρέπει τώρα να πούμε ότι το TPMS δεν θα κάνει τα πάντα, χρειαζόμαστε πιεσόμετρα ε, κατηγορίας 2. Μπορεί, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια καλή δικαιολογία. Να λέμε ότι τα συστήματα διαχείρισης στα αυτοκίνητα δεν θα είναι αρκετά αποτελεσματικά και χρειαζόμαστε ε, σε θέματα πιεσομέτρων ελαστικών. Αλλά δεν ακούσαμε πουθενά τέτοιο επιχείρημα. Οι εμπειρογνώμονες μας λένε ότι υπάρχουν ε, παράνομα ε, προϊόντα βάσει της οδηγίας. Θα δώσουμε όμως ε, κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θα τα καταστήσουμε παράνομα τα προϊόντα, μπορεί να δώσουμε και μία περίοδο 10 ετών ε, για την ε, απόσυρσή τους. Μπορεί να έχουμε μια διαδικασία phasing out. Λέμε ότι στη ψηφιακή τεχνολογία είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε μετρολογία. Ένα διεθνέ ε, πρότυπο συνήθω σα δίνει και ε, οδηγίες για το πώ να κάνετε την επισήμενση. Τα διεθνή πρότυπα δεν είναι ηλίθια. Ε, μπορείτε να το ζητήσετε αυτό. Οι επιρογνώμονές μα είναι όλοι μέλη του OML που είναι ο διεθνή οργανισμό Προτυποποίησης. Αυτοί είναι τα μέλη, οι δικοί μα επιρογνώμονες. Δεν είμαστε εμεί μέλο ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εμεί πάμε στι συνεδριάσει του, συζητάμε με του ρυθμιστέ, έχουμε επαφέ μαζί του, αλλά τα κράτη-μέλη είναι ε, αυτά τα οποία έχουν την διεθνή πρωτυποποίηση. Αν δεν μπορούν να γράψουν κάτι για τα διεθνή πρότυπα, ποιος μπορεί. Κατόπιν έχουμε μία ερώτηση για τις γλωσσικές απαιτήσει. Και η επισήμανση και οι απαιτήσει οι γλωσσικές κατά την άποψή μου δεν αποτελούν φραγμό για το εμπόριο. Τα ίδια λέει και ο ΠΟΕ. Κάποιος ρώτησε αν μπορούν να είναι υποχρεωτικά τα πρότυπα. Η απάντηση είναι όχι, δεν γίνεται, είναι θελοντικά. Είτε λοιπόν θα θεσπίσετε νομοθεσία, την οποία μπορείτε να τη θεσπίσετε χρησιμοποιώντα τα πρότυπα, αλλά εκεί αφού είναι νομοθεσία θα πρέπει να γράψετε πράγματα στην νομοθεσία που θα σας επιτρέπουν να αποφασίσετε. Μπορώ να δεχτώ ένα προϊόν ή όχι. Τα κράτη-μέλη όμως μπορούν κάλλιστα να το κάνουν αυτό, όπως και εμείς. Ακούσαμε και πολλές επικρίσεις γιατί δεν λάβαμε υπόψη την ε, προετοιμασία παραρτημάτων. Τον Απρίλιο του 2008 συγγνώμη, του 2007, τον Απρίλιο του 2007, είπαμε ότι θέλουμε να το δούμε από όλες τις πτυχές αυτό και για να, ανοίξουμε, να αφήσουμε κάποια ε, ενδεχόμενα ανοιχτά θα πρέπει να έχουμε παραρτήματα. Αν δεν το είχαμε πει αυτό, δεν θα είχαμε παράρτημα, θα έπρεπε να το ετοιμάσουμε την τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν ήταν λογικό να το πούμε στα κράτη-μέλη, αλλά ουσιαστικά η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έκανε υπόσχεση μετά να νομοθετήσει. Πάντα λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, αλλιώς δεν μπορούμε να νομοθετούμε, αλλά κάποιοι ε, δεν το κατανόησαν καλά και θεωρούν ότι έχουν ε, συνδρομή για την ε, νομοθεσία. Για κάποια κράτη-μέλη υπήρχε και ένα κίνητρο ότι δεν υπάρχει εντολή, τώρα ετοιμάζουμε και μια σχετική εντολή γι' αυτό. Για τη Γεωργία μιλήσαμε ήδη. Είπαμε ότι θα ήταν δύσκολο να αλλάξουμε τις συνήθειες ε, εκεί, γιατί τα πράγματα είναι ήδη εναρμονισμένα. Δεν ξέρω αν θέλουν περισσότερη εναρμόνιση στη Γεωργία. Δεν μας είπαν. Ε, τους ρωτήσαμε, μας είπαν δεν τη χρειάζονται. Ε, οι δεξαμενές πλοίων πρέπει να εναρμονιστούν για το διαμεθοριακό εμπόριο. Όχι, ε, δεν ε, υπάρχει θέμα εκεί μπορούν να περάσουν τα καράβια, είτε έχουν δεξαμενή είτε όχι. Αν θέλετε να έχετε διεθνή πρότυπα, κάντε στη χώρα σας ένα νόμο που θα βασίζεται στα διεθνή πρότυπα. There is a blocking, a blocking minority, yes, but uh, Μπορεί να υπάρχει και μία μειονότητα που θα ασκήσει βέτο, ναι, αλλά είναι λογικό να μην ακούσετε τα επιχειρήματα και της πλειοψηφίας. Το κατά πόσο θα αλλάξουμε την πρότασή μας, μας ρωτήσατε και αυτό, η απάντηση είναι εξ όσων γνωρίζω όχι, εκτός και αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Και ένας από αυτούς τους σοβαρούς λόγους που μας ε, παρουσιάστηκαν ήταν ότι θα υπάρχουν φραγμοί στο εμπόριο. Ρωτήσαμε τα κράτη-μέλη και δεν μας απάντησε κανείς κάτι τέτοιο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ε, δεν λάβαμε καμία νέα πληροφορία λοιπόν για προβλήματα, δεν λάβαμε καλές αιτιολογήσεις ε, από αυτά που έχουμε ακούσει στο Συμβούλιο. Όπως το βλέπουμε εμείς λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξανακάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου και να οπισθοδρομήσουμε, ε, διότι θα χρειαστούμε νέα ισχυρά επιχειρήματα. Ξοδέψαμε πάνω από μία ώρα για αυτές τις οδηγίες, τις οποίες θα να ξεκορτωθούμε κιόλας. Φανταστείτε πόσο χρόνο θα χρειαστούμε για να μιλήσουμε για οδηγίες που θέλουμε να κρατήσουμε και να ενδυναμώσουμε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, λέει ένας βουλευτής. Δεν θέλω να δημιουργήσω πρόσκομα στις εργασίες της Επιτροπής μας, ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά προσπαθώ να είμαι επικοδομητικός. Εξέτασα την ε, μελέτη επιπτώσεων, ακούσαμε και την παρουσίαση της Κομισιόν, αλλά δεν ακούσαμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Ε, υποβάλαμε διάφορα ερωτήματα που δεν μας απαντήθηκαν. Εγώ είχα πει ότι θα ήθελα στην μελέτη επιπτώσεων να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το πώς επηρεάζουν οι οδηγίες τα διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά δεν μου απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Ε, έχουμε μια πρόταση ε, της κυρίας Βάις Γκέρπερ για να συντάξουμε μια επιστολή. Ε, τι νομίζετε, έχουμε καμιά ελπίδα να λάβουμε και απάντηση. Αυτό είναι και ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει από αυτό. Ερωτήσεις, σχόλια. την υποστηρίζετε. Ωραία, μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν. Τώρα, να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, Solve It. Θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή, τον κύριο Μπουσόη, για να μας παρουσιάσει τις απόψεις του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να είμαι σύντομος. Θα πω δύο λόγια για το Solvit και μετά θα επισημάνω κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε κατά νου ε, λόγω της ε, προετοιμασίας και της εκθεσής μας. Όπως θα γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής μας, το Solvit είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη με στόχο να επιλύσουν προβλήματα τα οποία προκύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα κακής εφαρμογής ε, της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λίχτενστάιν, έχουν ε, συστήσει εθνικά κέντρα Solvit τις περισσότερες περιπτώσεις είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στο Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων. Τα κέντρα αυτά συνεργάζονται από κοινού μέσω μιας ε, ε, βάσης δεδομένων η οποία είναι online ε, για την επίλυση προβλημάτων τα οποία υποβάλλουν είτε πολίτες είτε εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. Ποιοι είναι οι κανόνες τώρα που διέπουν τις δραστηριότητες του Solvit. Πρώτον, έχουμε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2001, την οποία υιοθέτησε το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του. Επίσης, τα κέντρα Solvit ε, υιοθέτησαν ένα ε, κοινό σύστημα προτύπων και προδιαγραφών ε, το Δεκέμβριο του 2004 και το Solvit, να σας επισημάνω εδώ, τη λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2002. Το 2008 αυξήθηκε κατά 22% η ροή υποθέσεων του Solvit και για πρώτη φορά από τη δημιουργία του Solvit, όπως ε, σας είπα συστήθηκε τον Ιούλιο του 2002, είχαμε χίλιες υποθέσεις ε, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Solvit μέσα σε ένα χρόνο. Οι προσδοκίες για το 2008 είναι πολύ υψηλές, ε, το ποσοστό επίλυσης είναι περίπου της τάξης του 80%. Επιπλέον, το ποσοστό των υποθέσεων που επιλύονται μέσα στην προθεσμία των 10 εβδομάδων έπεσε από το 99% στο 74% το 2008, αλλά αυτό κυρίως ήταν λόγω έλλειψης προσωπικού. Θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο ποιοι είναι οι κύριοι τομείς ε, των υποθέσεων που επιλύθηκαν το 2008 και μετά θα περάσω στα σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη όταν θα ετοιμάσουμε την έκθεσή μας. Το πιο σημαντικό θέμα το οποίο αντιμετώπισε το Solvit ήταν θέματα κοινωνικής ασφάλισης, το, το 28%. Ένα 22% αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, ένα σημαντικό θέμα για τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως ακούσαμε και σήμερα το πρωί στις συζητήσεις ε, επί του θέματος. Η ελεύθερη μετακίνηση πολιτών και η νέα επικότητα είναι περίπου το 20% των υποθέσεων, κατόπιν φορολογία, εργασιακά δικαιώματα, ε, υπηρεσίες, εγκατάσταση, εγγραφή μοτοσυκλετών, πρόσβαση αγορά σε προϊόντα, άδειε οδήγηση, πρόσβαση σε εκπαίδευση, τελωνιακοί κανόνες και ε, συνοριακή έλεγχη. Αν λοιπόν θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα, νομίζω ότι το Solvit κάνει εξαιρετική δουλειά και προσεγγίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες της, ε, αποφεύγοντας ταυτόχρονα πολλά περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να καταλήξουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ε, προσφέροντας μία λύση με φιλικό τρόπο, ένα φιλικό διακανονισμό αν θέλετε, μέσω του δικτύου αυτό των κέντρων Solvit. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και να επισημάνουμε στην έκθεσή μας ε, κάποια σημαντικά στοιχεία για την εφαρμογή του Solvit. Καταρχάς, η έλλειψη προσωπικού, διότι σύμφωνα με την ίδια την έκθεση του Solvit ε, του 2008 πρόκειται για ένα πρόβλημα ε, που αφορά περίπου 10 χρόνια, χώρες. Συγγνώμη. Πρέπει επίσης να δούμε τις προδιαγραφές απόδοσης μεταξύ των κέντρων Solvit και των απαντήσεων που πρέπει να δίνονται, γιατί όλα αυτά γίνονται εθελούσιας βάσεως και δεν υπάρχει μία μεθοδολογία προσέγγισης. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε την καλύτερη ε, πληροφόρηση για την ύπαρξή τους καταρχάς και για τις δραστηριότητές τους κατά δεύτερον διότι επειδή δεν απασχολεί πολύ προσωπικό ε, το κέντρο Solvit και δεν υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν υπήρχε η δυνατότητα και οι ανθρώπινοι πόροι να ε, προβληθούν περισσότερο, να δημοσιοποιήσουν περισσότερο τις δραστηριότητές τους και να διασφαλίσουν ότι όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του δικτύου. Επίσης, θα πρέπει να συζητήσουμε στην έκθεσή μας το, την κακή εφαρμογή της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η προθεσμία των 10 εβδομάδων για τα Solvit για να επιληθεί το πρόβλημα ε, λειτουργεί καλά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της εσωτερικής αγοράς. Ε, οι υπηρεσίες βοήθειας για την ε, εσωτερική αγορά θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο στο Solvit Θα πρέπει και άλλες υπηρεσίες λοιπόν να συνδεθούν με αυτό το δίκτυο πιο επίσημα. Και θα πρέπει να επιλέγει με πιο συστηματικό τρόπο το Solvit ε, τις υποθέσεις που θα δεχτεί και τις υποθέσεις που θα απορρίψει με σαφή κριτήρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε δηλαδή μία μεθοδολογία σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να σταματήσω. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων αυτή για το Solvit. Με μεγάλη ανυπομονησία θα ακούσω τις απόψεις και τις προτάσεις των συναδέλφων και φυσικά και των σκιωδών εισηγητών. καθώς και όλων όσων εμπλέκονται στις δραστηριότητες του Solvit, που είναι τα άτομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσόη. Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Είναι ένας από τους πιο εργατικούς συναδέλφους και ένας που ασχολείται με πολύ άριθμες εκθέσεις. Τώρα, για αυτό το θέμα του Solvit. Φυσικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το Solvit. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει μια, να δοθεί μια άμεση βοήθεια στους ε, Ευρωπαίους πολίτες και να υλοποιηθεί στην πράξη η εσωτερική αγορά, αλλά το ποσοστό επιτυχίας ε, ποικίλει πολύ από κέντρο σε κέντρο. Γι' αυτό ακριβώς, νομίζω, θα έπρεπε να διερωτηθούμε ποιοι είναι οι λόγοι της ε, επιτυχίας ή της αποτυχίας των κέντρων Solvit. Τι εξηγεί τις διαφορές το διαφορετικό ποσοστό επιτυχίας από κέντρο σε κέντρο. Επίσης, οι επιχειρήσεις εκπροσωπούνται λιγότερο. Γι' αυτό θα πρέπει να επεκτείνουμε αυτό το σύστημα, θα πρέπει να δώσουμε στα κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι, γνωρίζει, ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο και ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Α, και θα πρέπει αυτό να γίνει και στα 27 κράτη-μέλη. Ε, ε, αυτό και θα έπρεπε να ε, στραφούμε με τα μηνύματα αυτά προς ε, το Διεθνές Επιμελητήριο. Διαπιστώνουμε όμως ότι υπάρχουν διάφοροι τομείς ε, οι οποίοι αναφέρονται σε δικαιώματα όπως η αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού και θα πρέπει να υπάρχει επικέντρωση στον τριμερή διάλογο διότι ε, υπάρχουν ορισμένες ε, καταστάσεις οι οποίες ε, μας θορυβούν και πολλές από αυτές δείχνουν ότι έχουμε λιγότερα περιστατικά από ό,τι στο παρελθόν όπως μέσω του διαδικτύου αλλά είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό θα έπρεπε να μπορέσουμε να διδαχθούμε από όλες αυτές τις πρακτικές διότι το κέντρο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Έχω εμπειρίες από την τσεχική δημοκρατία και το πιο βασικό είναι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Καταρχήν και ε, της δημοσίας διοικήσεως διότι αυτό εκδηλώνεται σε 38% των κέντρων και επιπλέον ο δημόσιος τομέας ε, κατά πάσα πιθανότητα δεν συνεργάζεται σωστά μαζί τους οπότε το Συμβούλιο και η Σουηδική Προεδρία θα έπρεπε να δώσει ένα σαφές μήνυμα στηρίξεως αυτών των κέντρων κατά τρόπον ώστε τα κράτη-μέλη και η δημόσια διοίκηση στα κράτη-μέλη αυτά να κινητοποιηθούν. Χαιρετίζω τις προτάσεις αυτές και συμφωνώ με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει παρουσιαστεί. η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή διότι πιστεύω ότι ο εισηγητής ε, έχει δώσει ένα σαφές μήνυμα πολύ ενθαρρυντικό διότι η, ε, όσον αφορά τα βοηθητικά θέματα είναι πολύ σημαντικά και θα έπρεπε να υπάρχει μία στενότερη συνεργασία ε, δηλαδή ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα των ε, περιορισμών ε, των δημοσιονομικών ε, των περικοπών διότι διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται καλύτερα σε ορισμένες χώρες από ό,τι σε άλλες οπότε καλό θα ήταν όλοι οι συνάδελφοι να έχουν υπόψη του το χρονοδιάγραμμα αλλά δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και τους ευχαριστώ πολύ για αυτά τα οποία ε, θέλησαν να μας επισημάνουν. Κυρία Ρίλε, θέλετε να πείτε κάτι. Ε, εδώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την πολιτική μας ομάδα γιατί δεν έχουμε αποφασίσει ποιος θα καταρτήσει την έκθεση, ίσως βρεθεί άλλο θέμα θύμα, αλλά ουσιαστικά ευχαριστώ τον εισηγητή, είναι θαυμάσιο θέμα και καλό είναι να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε ε, το θέμα αυτό στα κράτη-μέλη, ιδίω ε, την ανεπάρκεια προσωπικού, διότι θα πρέπει να πιέσουμε τις δικής των κρατών μελών, οι οποίες είναι υπεύθυνε και όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διεργασία θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την κυρία Ροϊτόβα για την πολύ καλά κατηρτισμένη έκθεση και έχω το συνέστημα ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε κάτι ακόμη σχετικά με το Solvit, ότι το Solvit είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το αμφισβητούμε και στις προηγούμενες, στα προηγούμενα χρόνια αντιληφθήκαμε ότι η συνειδητοποίηση ενισχύεται σε αυτό το πλαίσιο ε, της λύσεως δηλαδή των ε, διενέξεων χωρίς να καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το μηχανισμό του Σόλβι διότι σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχει δοθεί η αναγκαία σημασία στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με αυτή τη δυνατότητα επιλύσεως διαφορών. Ε, νομίζω ότι ο ρόλος ο δικός μας θα είναι να ενισχύσουμε αυτές τις ε, δραστηριότητες ενημερώσεως και διαδόσεως αυτού του εργαλείου διότι όταν όταν βλέπω ανθρώπους στην περιοχή μου, τους μιλώ για το Solvit και αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν γιατί μιλάμε. Και όταν αρχίζω να εξηγώ, αντιλαμβάνονται ότι είναι μια πολύ σημαντική δυνατότητα, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό και να το τονίσουμε στην έκθεση. Οπότε σας ευχαριστώ και ε, θέλω να ευχαριστήσω και για τη στενή συνεργασία. Ίσως καλό ε, θα ήταν αυτό να αναφερθεί ε, ε, στο την σελίδα μας. Η κυρία Γκέπχαρ τώρα. Όντως μπορεί να τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα του, της Επιτροπής μας διότι πολλοί απευθύνονται σε εμάς. Σε πολλές περιπτώσεις τους παραπέμπω στο Solvit και αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους. Οπότε για τους πολίτες νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουν οι ε, πολίτες ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και το λέγω για τον εξή λόγο διότι ε, τα κράτη δεν θέλουν να επενδύσουν όπως ε, τυχώς έχουμε διαπιστώσει και σε ταξίδια αποστολών ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ναι μεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται αλλά δεν, τα δεν χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν όλες αυτές τις εμπειρίες και έχουν δε ειδικευμένο προσωπικό το οποίο εργάζεται στον τομέα αυτό και γι' αυτό όπως είπε η κυρία Στάιλερ πρέπει να εξασκήσουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση κατά τρόπον ώστε η ε, πολίτες να ξέρουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Έχουμε έναν προπολογισμό και ίσως πρέπει να το θυμίσουμε στους πολίτες διότι στον προπολογισμό υπάρχει μία γραμμή του προπολογισμού και θα πρέπει στην Επιτροπή Προπολογισμού να φροντίσουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ε, προς αποφυγή μίας διαγραφής αυτής της γραμμής. Άρα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδοτήσεως μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να αναλάβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τέλος ε, Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα όσα άκουσα. Θυμάμαι ότι όταν ανοίξαμε το Solvit έγινε μία γιορτή. Και είχαμε πει τότε ότι έχουμε αυτό το θαυμάσιο εργαλείο ε, για το οποίο είναι περήφανα πολλά θεσμικά όργανα. Συχνά έχουμε εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους που δουλεύουν εκεί, ενώ από την άλλη έχουμε ε, επιχειρηματίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Solvit. Συχνά πηγαίνουν στο Solvit και φεύγουν απογοητευμένοι. Έχουμε λοιπόν αυτό το εργαλείο, να το χρησιμοποιούμε Όπω θα έπρεπε. Δεν χρησιμοποιείται επαρκώς. Δεν έχει αρκετά μέσα στη διάθεσή του και δεν είναι αρκετά γνωστό. Νομίζω ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κομισιόν, η Επιτροπή μας και όλοι μας είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε τον προπολογισμό. Πόσα μπορούν να δώσουν τα κράτη-μέλη στο Solvit και πώς θα προωθήσουμε αυτό το εργαλείο. Αυτά είναι τα στοιχεία και ελπίζω να υπάρξει και μια πολύ καλή συνεργασία και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα μπορούσαμε να τσεκάρουμε αυτή την πρόταση για το Facebook. Θα ακούσουμε και τη Ρία Γκρούμπερ από την Κομισιόν. Um, um, Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ε, ευρύτατη υποστήριξη που άκουσα σήμερα για το Solvit. Εμεί ε, πάντα υποστηρίζαμε στεναρά το Solvit και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην το υποστηρίζει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και είναι καλό νέο και για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το Solvit στα κράτη-μέλη. Ε, είναι δύσκολο πολλές φορές να πρέπει να πάνε στην πόρτα των άλλων Υπουργείων και να τους πούνε δεν εφαρμόζεται σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Φαντάζεστε ότι δεν τους αγαπούν και πολύ στα άλλα Υπουργεία ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αλλά κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά διότι διασφαλίζουν ότι όντως εφαρμόζεται ε, η νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς. Επομένως, αυτά τα νέα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, Εντό τη εβδομάδα θα υπάρξει ένα εργοστήριο για το ε, Solvit και θα πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του. Θα του τα δώσουμε τα νέα. Τώρα, είναι πολύ χρήσιμο να επισημάνουμε όλα τα θέματα τα οποία επισημάνουμε στην ετήσια έκθεση για τα τελευταία 7 χρόνια. Κάποια από αυτά τα θέματα έχουν παραμείνει προβλήματα και εσείς τα επισημάνατε όλα. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού στα κέντρα Solvit, διότι ε, ρωτήσαμε τα κέντρα Solvit και πάλι το Σεπτέμβριο τι γίνεται με το προσωπικό σας και πάλι όπως και τα προηγούμενα χρόνια το 1 τρίτο των κέντρων Solvit μας είπαν ότι δεν έχει επαρκές προσωπικό και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα χρήσιμο να το επισημάνετε κι εσείς στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Ένα ακόμα θέμα το οποίο τονίστηκε είναι το γεγονός ότι όλα τα κέντρα Solvit φαίνεται να κάνουν καλή δουλειά ως προς την προσέγγιση προς τους πολίτες, διότι οι υποθέσεις για τους πολίτες αυξάνεται. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ίδιο και για τις επιχειρήσεις. Αυτό επίσης ανακύπτει συνεχώς. Διαπιστώνουμε συνεχώς ότι ο αριθμός των ε, υποθέσεων από επιχειρήσεις στο Solvit μειώνεται. Φέτος χρησιμοποίησαμε το Standing Business Test ε, Panel για να βρούμε γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν το ε, Solvit και διαπιστώσαμε ότι δεν το γνωρίζουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν άλλους διάβλους για να προσεγγίσουμε και αυτούς τους χρήστες. Ε, τους ρωτήσαμε επίσης αν το γνωρίζατε το Silver θα το χρησιμοποιούσατε ή θα διστάζατε να το χρησιμοποιήσουμε. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας δισταχμός όταν το άκουσαν είπαν ότι θα το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν εξετάζουμε μια ε, στρατηγική καλύτερης προαγωγής για τις επιχειρήσεις. Θα το συζητήσουμε αργότερα εντός της εβδομάδας με τα κέντρα Solvit και θα σας ενημερώσουμε και εσάς για αυτά που έχουμε υπόψη. Τώρα για τον προϋπολογισμό. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υποστήριξη για το Solvit ε, και από πλευράς προϋπολογισμού. Αλλά το κονδύλιο που λαμβάνουμε από τον κοινοτικό προπολογισμό δεν είναι κονδύλιο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αυξήσουμε το προσωπικό στα κέντρα Solvit. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι προαγωγή του Solvit, να οργανώσουμε τα εργαστήρια, να διασφαλίσουμε ότι η βάση δεδομένων θα λειτουργεί και θα επικαιροποιείται όποτε είναι απαραίτητο, αλλά δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε το θέμα της έλλειψης του προσωπικού. Ένα ακόμα θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω, το οποίο ανέφερε και ο εισηγητής είναι το πρόγραμμα δράσης ε, για την ε, ε, συνδρομή στην ενιαία αγορά. Αυτό ξεκίνησε πέρσι και θέλουμε να συνδέσουμε πολύ καλύτερα όλες τις υπηρεσίες ενιαίας αγοράς και πολύ καλύτερα. Αυτό που κάναμε είναι να υπάρχει στενότερος σύνδεσμος μεταξύ της υπηρεσίας ε, πολιτών και των κέντρων Solvit ε, και γιατί ξέρετε ότι όταν έχετε ένα πολύ μικρό κέντρο και δεν υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη που ε, χρειάζεται για να απαντήσει στο ε, στο θέμα το οποίο του τίθεται μπορεί να αποτανθεί στην άλλη υπηρεσία και να λάβει τα στοιχεία που του λείπουν. Το δοκιμάσαμε πιλωτικά και είδαμε ότι λειτουργεί και τώρα θα το επεκτείνουμε και στα υπόλοιπα κέντρα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν και άλλα μέσα για να τους βοηθήσουμε λίγο με το θέμα της έλλειψης του προσωπικού. Τώρα, γιατί ο πρόγραμμα δράσης ε, για τη Single Market Assistance Services υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να προχωρήσουμε εκεί και θα θέλαμε να έχουμε ε, μία και μόνη είσοδο για αυτές τις υπηρεσίες ε, συνδρομής. Αυτή θα είναι η European Web δικτυακή πύλη, η οποία ελπίζω να είναι έτοιμη και προς το τέλος του έτους, ώστε να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε με το τι γίνεται με το πρόγραμμα δράσης, διότι έτσι θα μπορέσετε να έχετε και μια καλύτερη εικόνα του πώς το Solvit ταιριάζει σε αυτό το πρόγραμμα δράσης. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με τον εισηγητή να του δώσω όσες πληροφορίες χρειάζεται προκειμένου να ετοιμάσει την έκθεσή του. Συλλέγουμε και τα στατιστικά στοιχεία για την ετήσια έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί το Φεβρουάριο και θα δώσουμε τα στοιχεία και στον εισηγητή ώστε να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει για το σχέδιο έκθεσής του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκρούβερ. Ενθαρρύνω την Επιτροπή να το προωθήσει το Solvit, γιατί αν το χρησιμοποιούμε θα χαθεί. Αυτό ισχύει ό,τι τα χρησιμοποιείτε, καθίσατε ανώφελο. Αυτό ισχύει για πολλά πράγματα. Ο κ. Μπουσόη. Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν και δεν το λέω από ευγένεια γιατί οι ομιλητές ήταν γυναίκες, αλλά γιατί επί της ουσίας πιστεύω ότι υπάρχει μια θετική στάση, μια θετική ατμόσφαιρα εδώ για το Solvit και νομίζω ότι η έκθεση θα είναι θετική. Να σας προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα και να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι. Και εν συνεχεία θα εστιάσω σε δύο ε, σημεία τα οποία τα ανέφεραν πολλοί ομιλητές. Προτείνω λοιπόν μετά την ε, διαβούλευση με την Τζοάννα και τους υπαλλήλους της ΣΥΜΚΟ να έχουμε στις 5 Νοεμβρίου τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων να σταλούν στις 13 Νοεμβρίου τα κείμενα για τις μεταφράσεις στις 7 Δεκεμβρίου να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης ε, η προθεσμία για τις τροπολογίες να είναι λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα 11 Δεκεμβρίου στις 25 Ιανουαρίου ε, να δούμε τις τροπολογίες, να ψηφίσουμε στην ΙΜΚΟ τον Ιανουάριο και ε, στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου ή του Μαρτίου να ψηφίσουμε για την έκθεση. Ακούσαμε πολλά σημαντικά πράγματα, αλλά υπάρχουν δύο που είπαν πολύ, Καταρχάς το πρόβλημα της πρόθεσης. Το να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι αυτό το δίκτυο. Ομολογώ ότι πριν γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρότι ήμουν ε, Ρουμάνος βουλευτής, ε, δεν γνώριζα ότι υπήρχε το Σόρμπιτ. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Πολλοί πολίτες, πολλοί ε, επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν ακόμα την ύπαρξη του Solvit. Και πολλά από τα προβλήματά του μπορούν να επιληθούν από το Solvit. Προτείνουμε μια ξεχωριστή γραμμή του προπολογισμού. Στην Επιτροπή Προπολογισμών έχω την υποστήριξη πολλών συναδέλφων για να υπάρξει αυτή η χωριστή γραμμή του προπολογισμού. Φυσικά θα πρέπει να συζητηθεί και να τύχει διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Αλλά τουλάχιστον στην Επιτροπή Προπολογισμών ελπίζω η πρόταση αυτή να υιοθετηθεί. Αυτό ο προπολογισμό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόωθηση του δικτύου Solvit. Εν συνεχεία, δεύτερον, να πιέσουμε με την έκθεσή μα τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουμε να βοηθήσουν να επιληθεί το πρόβλημα της, του ανεπαρκούς προσωπικού και να προωθήσουν με τους πόρους που διαθέτουν, ε, να επανδρώσουν όλα τα κέντρα και στα 27 κράτη-μέλη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζομαι την συμβουλή τους, την υποστήριξή τους για να ετοιμάσω αυτή την έκθεση. Και σε ευχαριστώ που μου ξαναδώσατε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την ε, ακρίβεια που δείχνει η Επιτροπή μας, ε, με την τήρηση των προθεσμίων και των χρονοδιαγραμμάτων. Το επόμενο σημείο είναι το σημείο 13. Ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Κονιέτε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Κυρίες και κύριοι, υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν για το σχέδιο κανονισμού γιατί το θέμα είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τις υποδομές και σε ό,τι αφορά την ε, εσωτερική αγορά. Επίσης, άπτεται και της ε, ασφάλειας της Ευρώπης το θέμα αυτό. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για την ε, γρήγορη και επαγγελματική απόκριση ε, στην κρίση του Ιανουαρίου του 2009 και για το γεγονός ότι συνάφθηκαν τα σωστά συμπεράσματα από την κρίση. Τον Ιανουάριο του 2009 η κρίση απέδειξε ότι το θέμα της ασφάλειας του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο δεν μπορεί να επιληθεί σε επίπεδο κρατών μελών. Χρειάζεται κοινή δράση σε επίπεδο κοινότητας. και θα πρέπει να υπάρχει μια ε, ελεύθερη και σωστά λειτουργούσα ε, εσωτερική αγορά φυσικού αερίου με τη σωστή υποδομή. Όσο πιο ενσωματωμένη και ολοκληρωμένη είναι η υποδομή, τόσο πιο ε, βιώσιμη θα είναι οι μηχανισμοί της αγοράς και θα αντιστέκονται σε μακροχρόνιες διαταραχές. Θα ήθελα να συμπεριλάβω διάφορα θέματα στην ε, έκθεση, στην γνωμοδότηση. Καταρχάς, την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Εδώ υπάρχει μια πλειάδα ερωτημάτων, τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε. Καταρχάς, υπάρχει η μέγιστα, μέγιστη ευελιξία στους μηχανισμούς της αγοράς για να προσαρμόζονται στις διαταραχές αγοράς χωρίς παρέμβαση από τα κράτη-μέλη την κοινότητα. Υπάρχουν σαφή και επαρκή κριτήρια στον κανονισμό για την εισαγωγή κατεπηγόντων μέτρων εφόσον χρειάζονται αυτά. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχει επαρκή εξουσία η Κομισιόν για συντονισμό των δράσεων των αρχών των κρατών μελών για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τη εσωτερική αγορά σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα και αποτυχία στον ανεφοδιασμό τη εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να αφήσουμε μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη και στις εταιρείε φυσικού αερίου για να επιλέξουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ε, ανεφοδιασμού. Ή ίσως η έλλειψη σαφήνειας για τις δραστηριότητες των κρατών μελών και των εταιριών μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερους κινδύνους διαταραχής και περιπτώσει διαταραχής αγοράς. Θα ήθελα να σας πω ότι το πρότυπο ε, υποδομής νη 1 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να αμφισβητούμε την καθολικότητα αυτού του προτύπου, του νη 1, και το αν και κατά πόσον είναι κατάλληλο για τις διάφορες περιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Όμως είναι ένα βασικό μέτρο αναφοράς και βεβαίως οι ορισμοί και οι παράμετροι θα πρέπει να διευκρινιστούν σε σχέση με αυτό ε, και να διευκρινιστούν περαιτέρω. Ε, τώρα για την προστασία των καταναλωτών. Καταρχάς θα ήθελα να μιλήσω για τον ορισμό του προστατευόμενου καταναλωτή. Ίσως θα πρέπει να τους πούμε καλύτερα ε, χρήστες προτεραιότητας. το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να οριστεί με βάση τον συνολικότερο στόχο του κανονισμού και ίσως θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές. Επίσης, θα πρέπει να διερωτηθούμε γιατί ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής ε, αφήνει εκτός, ε, αφήνει μάλλον στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ε, τους πιθανούς χρήστες. Όταν μιλάμε για την προστασία των καταναλωτών, να μην ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για, για την ασφάλεια ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο και για τα μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση κρίσης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές να γνωρίζουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αρχών των κρατών μελών και των εταιριών παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση κρίσης. Και θα πρέπει να ενημερώνονται επίσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση κρίσης. Τώρα, ε, μία ερώτηση για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Οι πληροφορίες ε, που προβλέπει ότι θα παρέχονται ο κανονισμός είναι επαρκείς για να συντονιστούν οι δράσεις σε περίπτωση κρίσης. Και ιδίως αυτό αφορά τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών. Ή μάλλον τις αφορά, ερώτηση είναι και αφορά και τις συμφωνίες ε, παροχής με τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής φυσικού αερίου. Τέλος, κάτι για το κόστος. Τα μέτρα ασφάλειας του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο ε, συνεπιφέρουν μεγάλο κόστος. Φυσικά αυτό το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο από τις απώλειες που είχαν τα κράτη-μέλη σε περίπτωση κρίσης, όπου δεν υπήρχε κανένας κοινός ε, κοινοτικός μηχανισμός για την πρόληψη της κρίσης. Πιστεύω ότι το βάρος του κόστους θα πρέπει να πέφτει στους ώμους όλων ισότιμα. Και ο καονισμός θα πρέπει να είναι πιο σαφής και προβλέψιμος ε, και σε αυτό το τομέα επίσης. Τώρα, πώς θα εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη και τις κοινέ δράσεις των κρατών μελών στο μεταξύ. Φυσικά θα χρειαστεί πολύς χρόνος, ούτως ώστε τα μέτρα ε, που προτείνει ο κανονισμός να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί ο ίδιο ο κανονισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται σημαίνει ότι το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης θα είναι έτοιμο ε, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Εν συνεχεία, θα μπορούσαμε να έχουμε στην Επιτροπή μας τον Νοέμβριο την πρώτη ανάγνωση και να υιοθετήσουν τη γνωμοδότηση το Δεκέμβριο. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό και στενό, γι' αυτό καλώ όλου του συναδέλφου που θέλουν να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό αυτής της γνωμοδότησης να υποβάλουν τις προτάσεις τους τις επόμενες εβδομάδε, ούτω ώστε να μπορέσω να ετοιμάσω ένα σχέδιο γνωμοδότηση όσο πιο ευρύ και πλήρες γίνεται μέχρι τις 15 του μηνός. Είμαι νέα βουλευτής, νεοεκλεγήσα για την ακρίβεια και συνειδητοποιώ ότι πρέπει να μάθω πολλά. Αλλά γι' αυτό ακριβώς θα σας ήμουν ευγνώμων για οποιασδήποτε συνεισφορές ε, κατά την προετοιμασία αυτής της νομοδότησης. Ευχαριστώ κυρία Καλνιέτε. Φαντάζομαι ότι πολλοί θέλουν να βοηθήσουν αλλά εντυπωσιαστήκαμε με το καλό ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Ο κύριος Φιένικ θέλει να μιλήσει τώρα και μετά θα μπορέσουμε να δούμε μία παρουσίαση. Ευχαριστώ σε 15 λεπτά υπάρχει ψηφοφορία για το βραβείο Ζαχαρόφ και αυτό σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να παρουσιάσω τώρα την γνωμοδότηση των σοσιαλιστών και δημοκρατών επί του θέματος αυτού. Ε, ο κανονισμός αυτός είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας και εάν ε, διαβάσουμε προσεκτικά τι αναγράφεται ή την εισαγωγή θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε δύο θέματα. Καταρχήν τα προηγούμενα ε, έγγραφα επ' αυτού που αναφερόντουσαν ε, σε λιγότερο πολιτικά στοιχεία. Ξέρουμε τώρα ότι η πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ. Και ο, λόγος, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε το θέμα αυτό είναι ο ρυθμός αυξήσεως της κατανάλωσης του φυσικού αερίου. Είναι ένα είδος το οποίο είναι όλο και σε μεγαλύτερη ζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιτροπές οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν ε, επί του θέματος αυτού τεράστιος αριθμός και δεν με εκπλήσει γιατί πρόκειται για ένα πολύ ευρύ θέμα. Πρέπει όμως να παρακαλέσουμε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να γνωμοδοτήσει επίσης γιατί ε, είναι ένα θέμα που αναφέρεται στις ε, εξωτερικές σχέσεις. Είναι κάτι για το οποίο λοιπόν πρέπει και αυτή η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει. Μπορεί να είναι κάτι, ε, το στερεότυπο, αλλά ε, εμείς πρέπει να ε, ε, το εξετάσουμε από τη σκοπιά των καταναλωτών, της προσφοράς και της ζητήσεως. Και υπάρχουν τρία στοιχεία που μας επηρεάζουν. Καταρχήν, ο εισηγητής θα πρέπει να μπορεί να παραλαμβάνει την προμήθεια του φυσικού αερίου στην, στην ποσότητα που επιθυμεί και σε μία συμφέρουσα τιμή και νομίζω ότι ο τρόπος για την ε, ε, ρομήθεια ε, φυσικού αερίου είναι θέμα ζωής και θανάτου σε ορισμένες περι... περιπτώσεις. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό από πλευράς της ανθρώπινης ευημερίας, διότι τα θέματα ζωής και θανάτου είναι πολύ σημαντικά. Θα ήθελα όμως ε, εδώ να αναφερθώ στα θέματα που απασχολούν την πολιτική μου ομάδα, δηλαδή ε, τον προστατευόμενο χρήστη και τον προστατευόμενο λήπτη, ε, διότι μιλάμε για μεμονωμένους καταναλωτές, για σχολεία, για νοσοκομεία εδώ. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ορισμό πιο, ε, ε, ε, πιο εξεζητημένο για να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις και θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις ευθύνες διότι η ευθύνη αναλαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο στο οποίο το κράτος αναθέτει να εξασφαλίσει την ε, εγγύηση της προμήθειας τα, ε, οι προμήθειες πολλές φορές είναι σε χέρια ιδιωτών αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να είναι σαφές και ο κανονισμός αναφέρεται και στις προδιαγραφές προδιαγραφές ε, της ε, προσφοράς και της ε, των υποδομών. Αν λοιπόν αναφερόμαστε στην ε, παράδοση ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να παραλαμβάνει όσο φυσικό αέριο θέλει, χρειάζεται και υπάρχουν και δύο ακόμη θέματα επί των οποίων η πολιτική μου ομάδα έχουν ορισμένες επιφυλάξεις το άρθρο 7 σημείο 5 όπου λέγονται τα εξής. Η, η αρμόδια αρχή θα εγγυηθεί την ε, σωστή τιμή αγοράς και εδώ μιλάμε ε, ιδίω σε περιπτώσεις ε, καταστάσεως κρίσεως όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την προμήθεια του φυσικού αερίου και όπου προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον τελικό καταναλωτή, ιδίως όσον αφορά την τιμή, διότι ο τελικός καταναλωτής δεν επηρεάζει καθόλου την τιμή, ιδίως σε περίοδο κρίσεως. Ε, θα πρέπει λοιπόν κάπου να εμπλακεί. Και νομίζω ότι εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή να αναφερθεί το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα όμως πολύ να ακούσω τι έχουν να πούνε. Τέλος, ένα ακόμη θέμα που με απασχολεί είναι η ευθύνη του κράτους για να εξασφαλίσουμε το σωστό επίπεδο της βελτίστης προσφοράς. Μην ξεχνάμε τι έγινε στη Βουλγαρία, στα Βαλκα... στις Βαλκανικές χώρες, όπου υπήρξαν πολιτικά προβλήματα που διετάραξαν την προμήθεια του φυσικού αερίου και κάποιος πρέπει να αναλάβει τις ε, ευθύνες και να επιπληχθεί για την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας και να γνωρίζουμε ακριβώς ε, πόσο υπεύθυνο είναι ένα κράτο μέλος για την ε, παροχή φυσικού αερίου και πώς ένα κράτος μέλος μπορεί να βοηθήσει σε κατάσταση κρίσης. Είναι κάτι που πρέπει να καθορίσουμε. Το σχέδιο της, του κανονισμού είναι ένα καλό θέμα για να προωθήσουμε και θα πρέπει να ε, διαμορφώσουμε την πρότασή μας το ταχύτερο δυνατόν διότι ε, πλησιάζει ο χειμώνας και θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Ωραία. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον κύριο Βιενουά της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω την παρουσίαση αυτής της πρότασης, η οποία είναι πολύ σημαντική, λόγω και της ε, κρίσης τον Ιανουάριο. Είχαμε μια πολύ μεγάλη κρίση λοιπόν, όπου το 20% της ενέργειας ε, του αερίου που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν υπήρχε και υπήρχε και ευρωπαϊκή συνιστόσα διότι υπήρχαν αρκετές χώρες μόλι οι οποίες πλήττονταν απευθείας και πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πλήχθηκαν από αυτή την κρίση. Ουσιαστικά λοιπόν φαινόταν ότι η ε, κρίση θα πλήξει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά τη εσωτερική αγορά, νομίζω ότι ένα από τα καλά μαθήματα που πήραμε από αυτή την κρίση είναι ότι όντω η εσωτερική αγορά κατάφερε να λειτουργήσει και διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ροέ από δυσμά προ Ανατολά και διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν και ε, συμφωνίες φυσικού αερίου για να διασφαλίσουν ότι θα φτάσει το φυσικό αέριο σε αυτούς που πρέπει να φτάσει. Σε κάποιες χώρες διαπιστώσαμε ότι ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένα, υπήρχαν ε, ε, σχέδια κατεπίγουσας ανάγκης, υπήρχε και η ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου που είναι υπό την αιγίδα των κρατών μελών και του κλάδου του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορέσαμε να δούμε τι συμβαίνει και να λάβουμε και τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μετριαστούν τα προβλήματα. Επίσης, είδαμε και τα πιθανά ε, ωφέλη της ανάστροφης ροής, δηλαδή το να υπάρχει ένας αγωγός ο οποίος συνήθως λειτουργούσε από Ανατολή προς τη Δύση, να λειτουργεί πλέον προς ε, από τη Δύση προς την Ανατολή και προς το Βορρά και είχαμε και τη Βουλγαρία και την Ελλάδα εκεί στο τέλος της κρίσης. στη διάρκεια των ε, δύο εβδομάδων των περικοπών ε, έφτασαν ε, σε όλους το φυσικό αέριο, με εξαίρεση ίσως τη Βουλγαρία που ήταν η χώρα η οποία πλήχθηκε περισσότερο από την κρίση. Διαπιστώσαμε όμως ότι υπήρχαν και αρκετά προβλήματα και εδώ πρέπει να δράσουμε. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε απαραίτητη υποδημή για να φτάσει το φυσικό αέριο εκεί που απαιτείται, κυρίως από δυσμάς προς Ανατολάς έλλειψη προετοιμασίας κάποιων χωρών οι οποίες δεν ήταν ε, σε θέση να αντιμετωπίσουν την κρίση, ε, έλλειψη ανταλλαγής δεδομένων και έλλειψη διαφάνειας, καθώς επίσης και πλημελή διαμεθοριακό συντονισμό των κατεπηγόντων μέτρων, που σημαίνει ότι είχαμε μη παραγωγικά εθνικά μέτρα τα οποία έπληξαν κάποιες άλλες χώρες. Δεν υπήρχε αλληλεγγύη μεταξύ χωρών μελών διότι δεν δημιουργείται η αλληλεγγύη εν μία νυχτή ειδικά σε περίοδο κρίσης και φυσικά δεν υπήρχε και κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου που σημαίνει ότι δεν ήμασταν και κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ο κανονισμός τώρα βασίζεται στο άρθρο 95, κοινά προδιαγραφές για την ασφάλεια εφοδιασμού και είναι ε, ε, ένα άρθρο το οποίο αφορά στην νέα αγορά. Είναι ζωτική σημασία να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ροή φυσικού αερίου μέσω μιας καλά λειτουργούσα εσωτερικής αγοράς και αυτό για να αποφύγουμε και στρεβλώσεις της αγοράς στη διάρκεια κρίσεως και ταυτόχρονα η αγορά να μπορεί να λειτουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να φτάνει το φυσικό αέριο σε όλους τους πελάτες. Το βασικό όμως μάθημα ε, του Ιανουαρίου είναι ότι η καλύτερη διασφάλιση για την ασφάλεια εφοδιασμού είναι η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πολύ καλά. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κίνητρα για να επενδύσουμε σε υποδομές όπου αυτές δεν υπάρχουν και επίσης ε, ενσωματώσαμε αυτόν τον κανονισμό στο προσφάτως υιοθετημένο τρίτο πακέτο εσωτερικής αγοράς. Έχουμε τον κανόνα, ε, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη συνεργασία των ε, ρυθμιστών ενέργειας, καθώς επίσης και την ενίσχυση της συντονιστικής ομάδας στον τομέα του φυσικού αερίου. Και φυσικά αυτοί οι δύο νέοι φορείς θέλουμε να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου που ε, υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τρίτο πακέτο θα προσφέρει περισσότερη διαφάνεια για το δίκτυο και κυρίως τη χρήση του δικτύου. Ο στόχος λοιπόν του κανονισμού είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη προστασία των πελατών φυσικού αερίου ε, σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που είπε και ο τελευταίος ομιλητής, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει φυσικό αέριο στους πελάτες. Και εδώ χρειαζόμαστε κοινέ προσδιογραφέ ε, για προστασία, για παροχή στους προστατευόμενους πελάτες, που είναι δηλαδή τα νοικοκυριά, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν φυσικό αέριο και σε περίπτωση κρίσης. Βέβαια, αν θέλετε να το κάνετε αυτό, σαφώς θα πρέπει να υπάρχει και καλύτερη πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα αποδεκτό ε, κοινό επίπεδο ετοιμότητας ε, και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό ίσως επίπεδο που είναι πολύ σημαντικό. Η περιφερειακή συνιστόσα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για το θέμα αυτό διότι ένα κράτος μέλος μπορεί να μην μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά όλους τους κινδύνους, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε με συντονισμένο τρόπο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και αυτό είναι και το στοιχείο της αλληλεγγύης, το οποίο θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα. Φυσικά η διαφάνεια είναι προαπαιτούμενο για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσεως. Ο κανονισμός στην πράξη χρησιμοποιεί ένα νέο βασικό στοιχείο, το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει μία αξιολόγηση κινδύνου που βασίζεται σε δύο σε προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία προδιαγραφή υποδομής, την 1 και δύο προδιαγραφές εφοδιασμό για τους προστατευόμενους πελάτες, που είναι 7 ε, ημέρες ε, για, την, ε, για τις περιόδους εχμής του χειμώνα και 60 ημέρες για την υψηλή περίοδο εχμής. Και αυτό φυσικά μας οδηγεί και σε προγράμματα δράσης προληπτικά και κατεπήγοντα προγράμματα για την αντιμετώπιση. Έχουμε τρία επίπεδα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό όμως και περιφερειακό επίπεδο, θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, αν δούμε το δίκτυο νήμιον 1, ο οποίος είναι ο δίκτυς ε, της υποδομής. Τι συμβαίνει αν η βασική σας υποδομή έχει πρόβλημα. Υπάρχουν ε, αρκετές άλλες υποδομές ή αρκετά άλλα μέσα για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν είναι τόσο καλά ε, προετοιμασμένες και υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες ε, διαθέτουν υποδομή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να δούμε και αυτό το δίκτυο με μια κάποια ευελιξία, να δούμε όλη την υποδομή, όχι μόνο τους αγωγούς, αλλά και τις δυνατότητες αποθήκευσης, ε, σταθμούς ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου, δυνατότητα αποθεματικού και όλους αυτούς που έχουν θέματα προστασίας. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια αξιολόγηση κινδύνου που θα βασίζονται σε αυτό το βασικό δίκτυ, διότι είναι βασικό στοιχείο της ευθύνη που πρέπει να φέρει κάθε κράτος μέλος στο σύστημα. Ξέρετε ότι ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος κάποιες χώρες να μην μπορούν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και να βασίζονται στις γείτονες χώρες νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτές τις μορφές τα προβλήματα και να διασφαλίσουμε ότι κάθε κράτος μέλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και από εκεί και πέρα να προκύψει ο μηχανισμός της αλληλεγγύης επί τη βάση της εμπιστοσύνης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κοινοτική συνιστόσα τώρα θα ήταν ουσιαστικά ότι η διαδικασία της ανάλυσης κινδύνου και η εκπόνηση προγραμμάτων δράσης και κατεπηγόντων προγραμμάτων θα πρέπει να την χάνει κάποιες καθοδήγησεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή που θα καθοδηγεί και θα πρέπει να πιέζει τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που μπορεί να είναι και ο περιφερειακός τρόπος. η Κομισιόν ε, μπορεί και να συστήσει να υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα όπου θεωρεί ότι υπάρχουν ωφέλη εξ αυτού. Επίσης, θα θέλαμε να ενισχύσουμε το ρόλο της συντονιστικής ομάδας φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, θα ε, πρέπει να έχουμε συνεργασία και με την υπηρεσία με τους ρυθμιστές της ενέργειας και με την Enso Gas. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα η Κομισιόν να ζητήσει από κάποιο κράτος μέλος να αποφύγουν να λάβουν ε, μέτρα ε, κατά κάποιο άλλο κράτος μέλους. Ε, αυτό είναι μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά πιστεύουμε ότι σε περίπτωση κρίσης να μπορεί ένα κράτος μέλος να μην λάβει μέτρα τα οποία μπορεί να είναι αντιπαραγωγικά για κάποιο άλλο κράτος μέλος. Και φυσικά όλα αυτά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε αυξημένη διαφάνεια της αγοράς φυσικού αερίου εν γέννη και κυρίως σε περίοδους κρίσης. Αυτά λοιπόν είναι τα όσα αφορούν στο υπέβαθρο αυτού του κανονισμού και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εγώ να κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα α, προβλήματος. Μπορείτε να μου πείτε ένα, ενίδη παραδείγματος, εθνικό μέτρο που να είναι αντιπαραγωγικό. Υπάρχουν δύο είδη μέτρων. Καταρχάς να πούμε ότι όλο το αποθεματικό πηγαίνει για, εθνικούς, για εθνική χρήση. Ε, τα αποθεματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διασυνοριακά και να παγώσουμε τη χρήση του αποθεματικού δεν είναι ένα καλό μέτρο βέβαια, δεν είναι ιδανικό μέτρο. Επίσης, το να συνδέσουμε κάποια μέτρα τα οποία έχουν στρεβλωτικό χαρακτήρα στην αγορά, που μπορούν να βελτιστοποιούν, ας πούμε, τις εισαγωγές και να δώσουμε ένα μήνυμα στους operator ότι δεν θα πρέπει να εξάγουν σε χώρες που χρειάζονται όμως ε, το φυσικό αέριο. Τέτοιου τύπου μέτρα μπορούν να δημιουργήσουν ε, προβλήματα και να έρθουν σε αντίφαση με το στόχο της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν ερωτήσεις από την Επιτροπή, από τα μέλη της Επιτροπής. Κυρία Κονιέτε, έχει ξανά το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίασή της. Είμαι έτοιμη να συνεργαστώ στενά με όλες τις ομάδες και με όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό. Θα ήθελα να συναντηθώ λοιπόν με τους σκιώδεις εισηγητές το συντομότερο δυνατόν. Πάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 14, που είναι η παρουσίαση της μελέτης για την αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιάννη Σίλβε. And uh, multi-talent expert. είσαστε εμπειρογνώματος με πολλά ταλέντα. Καλώς ήλθατε. Πάλι έχουμε παρουσίαση PowerPoint. Move. Thank you, Madam Chairman. I'm happy to be back. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Ε, σήμερα το πρωί έκανα πάλι μια παρουσίαση για όσους δεν ήσασταν, το λέω. Μας ζήτησαν να κάνουμε μια μελέτη που αξιολογεί την ε, εποπτεία της αγοράς, όπως ε, προβλέπεται στα κράτη-μέλη. Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι να κάνει μια επισκόπηση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα κράτη-μέλη για να ενδυναμώσουν τα μέσα και τους φορείς εποπτείας της αγοράς. Και είναι βέβαια τμήματα του πακέτου αγαθών που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2008. Ε, αυτό που εξετάζουμε σε αυτή τη μελέτη είναι ποια μέτρα έχουν ληφθεί από τα κράτη-μέλη για την αποτελεσματική λειτουργία και την ενδυνάμωση της ε, εποπτείας της ε, αγοράς ε, και τους πόρους που έχουν ε, προβλέψει τα κράτη-μέλη γι' αυτό. Κοιτάμε τα προγράμματα εποπτείας της αγοράς ε, που έχουν προωθήσει τα κράτη-μέλη και επίσης πόσα προϊόντα έχουν ανακαλυφθεί ότι παρουσιάζουν σοβαρό το κίνδυνο και τι μέτρα έχουν ληφθεί για να ανοιχνευθούν. Και επίσης μιλάμε για την εγκατάσταση, την ε, θέσπιση των ε, μηχανισμών ελέγχου στα κρατη πάντα με βάση τον κανονισμό. Το σημείο φετηρίας λοιπόν είναι το πακέτο αγαθών και πιο συγκεκριμένα ένας από τους ε, κανονισμούς ο 1765. Το πακέτο για τα αγαθά έχει σκοπό να εξασφαλίσει ένα κοινό πλαίσιο για τη βελτίωση της υποδομής εποπτείας της αγοράς. Ε, δίνει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ε, θέση σε εμπορία των προϊόντων. Ο συγκεκριμένος κανονισμός που εξετάζουμε είναι τμήμα του πακέτου αγαθών, όπως σας είπα, και εισάγει κάποιες διατάξεις για την πιστοποίηση και την εποπτεία της αγοράς. Θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2010 και τα κράτη-μέλη αναμένεται να έχουν ήδη λάβει τα μέτρα για να ενδυναμώσουν την εποπτεία της αγοράς. Ιδίως γιατί ο κανονισμός προβλέπει μια αυξανόμενη ευθύνη για τις ε, αρχές των κρατών μελών. Αυξανόμενη ευθύνη. Παραδείγματο χάρη την απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων ε, από την αγορά και την καταστροφή τους, αν Για αυτή τη μελέτη έχουμε έρθει σε επαφή με εκπροσώπου όλων των κρατών μελών και επομένω έχουμε μια υποπτική εικόνα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ενδελεχή γνώση του πώς λειτουργούν τα διάφορα κράτη-μέλη για τις, ε, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας αγοράς. Έχουμε επιλέξει 7 χώρες που χρησιμοποιούμε Χρησιμοποίησαμε δηλαδή νέα κράτη-μέλη, παλιά κράτη-μέλη, μεγάλα κράτη-μέλη, μικρά κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη, έχουμε δει ποιο έχει συγκεντρωτική ε, προσέγγιση, ποιο αποκεντρωμένη, το επίπεδο συνεργασία των κρατών μελών και ειδικέ ανάγκε. Παραδείγματο χάρη, κάποιε χώρε, ε, όπω το Ρότερνταμ και το Αμβούργο, ε, λαμβάνουν πολλές εισαγωγέ, ας πούμε, γιατί περνάνε πάρα πολλά αγαθά ε, μέσα από αυτά τα λιμάνια. Η Γερμανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Λετωνία είναι χώρε που επιλέξαμε για να μελετήσουμε. Τα πορίσματα της μελέτης. Καταρχάς, Κοιτάμε τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τη λειτουργία και την ενδυνάμωση των αρχών εποπτείας της αγοράς. Κοιτάξαμε τι πόρους έχουν δοθεί σε αυτές τις αρχές εποπτείας της αγοράς και βρήκαμε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία του στα κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει περισσότερους ανθρώπινους ή οικονομικούς πόρους σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για αυτόν τον λόγο. Καταρχάς, ε, πολλές χώρες ε, έχουν γονατίσει κάτω από την ε, πρόσφατη κρίση και επομένως έχουμε μειώσεις περικοπές στο δημόσιο τομέα, σε πολλούς τομείς και στην εποπτεία της αγοράς. Ενώ άλλες χώρες έχουν ήδη ένα σύστημα εποπτείας αγοράς που συμμορφώνεται με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός ή με μικρές αλλαγές θα συμμορφωθεί. Και επομένως δεν χρειάζονται ή δεν θεωρούν ότι χρειάζονται να προσθέσουν ε, πόρους ε, στο σύστημά τους. Αυτή είναι η βασική λόγη λοιπόν, γιατί στις περισσότερες χώρες ε, οι πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί είναι περίπου ίδιοι. Μεταξύ των κρατών μελών που έχουν πόρους, επαρκείς πόρους για την εποπτεία της αγοράς, έχουμε τη Σουηδία, που είναι μια χώρα καλών πρακτικών, που συντονίζει αποτελεσματικά τις δραστηριότητε των αρχών εποπτείας αγοράς μέσω ένας, ενός συμβουλίου που συντονίζει αυτές τις δραστηριότητες. Ένα άλλο παράδειγμα καλής και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων είναι η βαλτική συνεργασία που ξεκινάει από τη Γερμανία και το λιμάνι του Αμβούργου και εμπλέκει διάφορα κράτη-μέλη, ιδίως τα νέα κράτη-μέλη που έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσει. Τα κράτη-μέλη, με βάση το άρθρο 18 του νέου κανονισμού, πρέπει να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς που θα περιγράφει τις δραστηριότητες, τις αρχές που εφαρμόσουν κτλ. Από τα κράτη-μέλη που έχουν ξεκινήσει τη σύνταξη ενός προγράμματος, είναι η πλειοψηφία. 18 κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει. Μιλάμε για νομικές δομές, διοικητικές δομές, ε, έχουν ψάξει να δουν αν θα έχουν ε, συγκεντρωτική προσέγγιση ή περιφερειακή προσέγγιση. Ένα από τα σημεία που βρήκαμε είναι ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει περιφερειακή προσέγγιση, παραδείγματος χάρη στα ομοσπονδιακά κράτη, Χρειάζεται παρόλα αυτά εθνικό συντονισμό. Ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια κοινή εθνική προσέγγιση για την εποπτεία της αγοράς. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει βέλτιστος τρόπος ε, τομεακός, εθνικός ή περιφερειακός, γιατί εξαρτάται από την ε, φύση και τη λειτουργία της αγοράς της κάθε χώρας. Κάθε χώρα λοιπόν θα πρέπει να επιλέξει την προσέγγιση που τη ταιριάζει καλύτερα. Επίση, βρήκαμε ότι οι νέα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει την ε, δημιουργία προγραμμάτων εποπτείας της αγοράς. Οι λόγοι είναι μεικτοί. Ένας λόγος είναι ότι δεν έχουν αρκετή εμπειρία σύνταξη τέτοιων προγραμμάτων και δεν έχουν καμία βεβαιότητα για το πώς θα πρέπει να κινηθούν. Κάποιες άλλες χώρες έχουν περιορισμένους πόρους στη διάθεσή τους και ε, σε ορισμένε περιπτώσεις είναι αμφισβητούσιμο το αν θα, αμφισβητήσιμο το αν θα έχουν εποπτεία της αγοράς ή αν θα πρέπει να ξοδέψουν τους ελεύθερους πόρους για τη σύνταξη των προγραμμάτων. Οι χώρες αυτές λένε ότι θα ήθελαν ε, να του δοθούν περισσότερε κατευθύνσει και κατευθυντήριες γραμμέ από την Κομισιόν για το πώ θα πρέπει να κινηθούν και να συντάξουν αυτά τα προγράμματα, ποια θα πρέπει να είναι η δομή, τι είδου πληροφορίε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτά τα προγράμματα κτλ. Η αντίδραση τη Κομισιόν ήταν ότι δεν περίμεναν ότι χρειάζονταν κάποια κράτη τόση μεγάλη υποστήριξη. Δεν περίμενε η Κομισιόν. Ίσως όμως είναι καλό που υπάρχει αυτή η ανάγκη για καθοδήγηση για να υπάρχει όχι ακριβώ μια εναρμονισμένη προσέγγιση, γιατί είναι υπερβολικός όρο, αλλά να υπάρχει ένας κάποιο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή να μιλάνε τα ίδια θέματα στα προγράμματά τους και να προωθούν τα ίδια θέματα μέσω των προγραμμάτων τους. Όσον αφορά τα, τον αριθμό των προγραμμάτων τα οποία ευρέθηκαν, ε, υπάρχουν ε, διάφοροι κίνδυνοι και μία από τις βασικές ε, πηγές πληροφοριών είναι το σύστημα RAPEX το οποίο αναφέρεται σε όλα τα, προϊόντα τα οποία έχουν διαπιστωθεί και όσον αφορά το RAPEX υπήρξε μία σαφής αύξηση ε, των ε, κοινοποιήσεων την τελευταία πέντα ετία ενώ σαν αφορά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ε, παρουσιάστηκε μία μείωση όσον αφορά τις κοινοποίησεις των μελών. Το RAPEX μπορεί να θεωρηθεί επιτυχές και αυτό οφείλεται εις την, ε, ε, ε, το ότι επικεντρώθηκε στα παιχνίδια μετά από το σκάνδαλο της Ματέλ για τον αριθμό των επικινδύνων παιχνιδιών και ένα μεγάλο ποσοστό των κοινοποιήσεων οφείλεται στα παιχνίδια βεβαίως υπάρχουν και πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών όπου επίσης ε, ζητείτε να υπάρξει ε, μία ε, μία ενημέρωση για τα διάφορα προϊόντα. Έπρεπε επίσης ε, να έρθει κανείς ε, σε επαφή με τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών όπου δεν αναμένεται μία αύξηση διότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και υποτίθεται ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει ένας ίσος αριθμός κοινοποιήσεων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι παρόλο που έχουμε το RAPEX υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί ε, μεταξύ των οποίων ο πιο βασικός είναι ότι ε, δεν υπάρχει ένας ορισμός του τι σημαίνει ένα επικίνδυνο προϊόν, δηλαδή πόσο επικίνδυνο πρέπει να είναι για να ε, κοινοποιηθεί και υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές στα κράτη-μέλη όσον αφορά το τι αναφέρουν και πώς το αναφέρουν. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα καλό σύστημα για να συγκρίνουμε τις πληροφορίες, αλλά τώρα με τους περιορισμούς τους το RAPEX θεωρείται το καλύτερο σύστημα και σε σχέση με τις άλλες βάσεις δεδομένων που αναφέρονται εις ε, τα τρόφιμα στις ζωοτροφές και ε, στον πίνα βαθμολογήσεως των προϊόντων έχουμε τα πιο καλά αποτελέσματα. Μετά εξετάσαμε την κατάρτιση των συστημάτων ελέγχου και τα διάφορα συστήματα ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι στις χώρες όπου υπάρχουν συστήματα για συνεργασία σε εθνικό επίπεδο όπως η Γερμανία και η Σουηδία ε, παρόλο που τα συστήματα είναι αρκετά αποκεντρωμένα με διάφορες ε, αρχές εποπτείες της αγοράς οι ε, αρχές αυτές ε, Αλλά ενημερώνονται για τα προϊόντα και την πορεία τους ε, ενώ ε, ορισμένες πρακτικές έχουν επίσης προωθηθεί σε πολλά κράτη τα οποία καταγράφουν και διανύμουν τα προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτηρίσει ως επικίνδυνα. Η ε, Σουηδία έχει ε, ένα θαυμάσιο σύστημα ε, συντονισμού μεταξύ των αρχών οπότε δεν έχει ακόμη αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα για διασυνοριακές ανταλλαγές. Προηγουμένως ανέφερα την συνεργασία της Βαλτικής. Ο γερμανικός, το γερμανικό λιμάνι του Αμβούργου είναι το κέντρο για αυτήν την συνεργασία της Βαλτικής όπου διάφορες χώρες ε, ε, ε, αλληνοενημερώνονται για τις πληροφορίες και για τα προϊόντα που διέρχονται από το λιμάνι του Αμβούργου και προχωρούν σε άλλες χώρες και τώρα αυτή η συνεργασία επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές που δεν έχουν καμία σχέση με τη Βαλτική όπως παραδείγματο χάρη η Κροατία η οποία έχει ε, εξελιχθεί σε μια σημαντική ε, χώρα ε, ενημέρωσης για να γνωρίζει κανείς τι γίνεται. Uh, ένα άλλο βασικό σύστημα το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι η Ολλανδία η οποία χρησιμοποιεί μια στρατηγική αξιολόγησης κινδύνου για να καταρτήσει προτεραιότητες μέσω του μεγάλου λιμανιού του Ρότερνταμ όπου διέρχονται τεράστιες ποσότητες ε, αγαθών δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλα. Χρησιμοποιούν λοιπόν μια στρατηγική αξιολόγηση του κινδύνου εξετάζοντας τι είδη προϊόντος ή από ποια χώρα προελεύσεως ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα και εστιάζοντας τις προσπάθειές τους σε αυτά τα προβλήματα, τα, ε, προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να εντοπίσουν τα προϊόντα ε, πριν καταλήξουν στην αγορά, ενώ σε άλλες ε, χώρες ε, τα προϊόντα εντοπίζονται όταν ε, έχουν πια φτάσει στην αγορά και έχουν εντοπιστεί από τους καταναλωτές. Είναι λοιπόν ένας ε, τρόπος για να παρουσιαστεί αυτό το σύστημα και να προωθηθεί και ε, να ενημερωθούν και ε, χώρες οι οποίες έχουν δημοσιονομικούς περιορισμούς και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιλέξουν καλύτερα ε, ποια προϊόντα θα ελέγξουν. Τα περισσότερα προϊόντα αναφέρονται σε ένα σύστημα πιο δραστικό παρά κατασταλτικό Δηλαδή, σε ορισμένες χώρες το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά, αλλά υπάρχει πρόβλημα όπου υπάρχει χαμηλός δείκτης εμπιστοσύνης των πολιτών. Παραδείγματος χάνει στη Βουλγαρία όπου υπάρχει χαμηλός δείκτης εμπιστοσύνης των πολιτών, δεν κάνουν καν τον, τον κόπο να ενημερώσουν τις αρχές για τα επικίνδυνα προϊόντα. Δηλαδή εκεί στη Βουλγαρία οι ε, σύνδεσμοι βιομηχανιών δεν ε, ε, δίδουν πολλές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων για λόγους λένε ανταγωνισμού και χρειάζεται να καταναλωθούν πολύ μεγαλύτερα ποσά για να διαπιστωθούν ποια προϊόντα είναι επικίνδυνα. Συνοψίζοντας λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει η στρατηγική αυτή αξιολογήσεως του κινδύνου για τα προϊόντα προτού καταλήξουν στην αγορά και υπάρχει ένα συμβούλιο εποπτείας της αγοράς το οποίο λειτουργεί με αποκεντρωμένη μορφή και συνεργασία για να υπάρξει συνεργασία όπως στα πλαίσια της συνεργασίας της Βαλτικής. Υπάρχουν δηλαδή τρία στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους συνδυασμούς κατά τρόπον ώστε να διεξαχθούν να διεξαχθούν οι ε, έλεγχοι αυτοί με χαμηλό κόστος και αποτελεσματικά και με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών. Ευχαριστώ και αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Ευχαριστώ κυρία Σίλβερ. Members wishing to... Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να θέσει κάποια ερώτηση, να σχολιάσει. Ο κύριος Κότσμαν πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην πρακτική μου, επειδή είμαι ε, ε, ε, βουλευτής στο προϊόν του κρατηδίου μου έχω συνηθίσει να κάνουμε ερωτήσεις και να ελέγχουμε τα προϊόντα στα σύνορα. Δηλαδή όταν φτάνει ε, το προϊόν από την Κίνα π.χ. στη Γερμανία και υπάρχει μια αποκέντρωση ε, για τα κρατηδία στη Γερμανία οπότε μπορεί κανείς να επέμβει ακόμη και σε ένα λιμάνι κάνει σαν το Ρότερνταμ παραδείγματο χάρη, αλλά είναι πιο δύσκολο διότι ε, πρέπει κανείς ε, να ελέγξει ε, γιατί παραδείγματο χάρη ένα παιχνίδι πολλές ε, φορές ε, ε, δεν μπορεί όπως και άλλα προϊόντα να εισαχθεί χωρίς τη συνένεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οπότε παραδείγματος χάρη στο Ρότερνταμ υπάρχει ένα ε, ε, πρώτο σταθμός, παρακολουθούμε δηλαδή και την εσωτερική διακίνηση ε, στις ποτάμιες οδούς, γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε από τα κρατήδια να επέμβουν μόνο όταν θα έχει το προϊόν εισαχθεί στη χώρα. Οπότε πέραν αυτού η Υπάρχει επίσης ε, η δυνατότητα να επέμβει κανείς περισσότερο στα λιμάνια με μια αρχή αλληλεγγύης χωρίς δηλαδή ε, να ε, δοθούν ειδικέ αρμοδιότητες σε κάθε κρατήδιο αλλά στα εξωτερικά σύνορα στην Ιταλία παραδείγματος χάρη ενδέχεται να μην υπάρχει αποδοχή και αν χρειαστεί εκεί ε, να γίνουν τα, οι έλεγχοι εφόσον το προϊόν έχει ήδη ισχύσει, ε, εισέλθει στην Ευρώπη τότε πολλά κράτη θεωρούν ότι ήδη έχει υπάρξει ένας πρώτος έλεγχος και δεν υπάρχει άλλη εποπτεία σε χώρες όπως είναι η Γερμανία παραδείγματο χάρη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ισχύσει η ε, η ε, αλληλεγγύη στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και στους, στα σημεία εισόδου ώστε να μην χρειαστεί μετά να επιδιορθώνουμε τα κακό κείμενα. Θα ήθελα να πω ότι ούτως ή άλλως η αρχή και το τέλος κάθε ρυθμίσεως είναι να γίνονται σεβαστές. Δεν πρέπει δηλαδή να βασιστεί κανείς στο ότι υπάρχει ένας κανονισμός και ακόμη και αν δεν γίνει σεβαστός να θεωρήσουμε ότι η κυρία, Η Στάιλερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Λυπάμαι που δεν έχουμε άλλα μέλη εδώ, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά που επισημάνατε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και η ανάλυση σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να ακούσω κάποια πράγματα για τα συμπεράσματά σας. Είπατε τα κράτη-μέλη δεν ε, διαθέτουν κονδύλια ή ανθρώπινο δυναμικό ε, στην εποπτεία της αγοράς. Αναφερθήκατε και στην οικονομική κρίση και παρατήρησα ότι αν δείτε στο παράρτημα έχουμε κάθε κράτος ε, μέλος, τη σελίδα 44-45, και παρά το γεγονό ότι όλοι λένε, όχι όλοι, αλλά η Ελλάδα λέει όχι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια περίεργη διαδικασία συντονισμού ad hoc. Μήπως μπορείτε να μα εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει. Νομίζω ότι η μόνη χώρα που δεν έχει φορέα συντονισμού είναι η Ελλάδα. Αυτή η περιγραφή ad hoc λοιπόν θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Στα κράτη-μέλη Όσον αφορά στο συντονισμό, βλέπουμε ότι μόνο η Κύπρος και η Δανία λένε ναι και μόνο η Γερμανία λένε ότι θα πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι. Περιγράψατε και την αύξηση στη διάρκεια μιας πενταετίας των επικίνδυνων προϊόντων που διαπιστώνονται, παρά το γεγονός ε, ε, ότι λέτε ότι κυρίως αφορούν σε παιχνίδια, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα θέματα απασχολούν τους καταναλωτές και αν ο βασικός μας ε, στόχος είναι η προστασία του καταναλωτή, το θέμα του πώς λειτουργεί η εποπτεία είναι σημαντικό. Αυτό που είπε ο προλαλής σας είναι πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι από τους πολύ μεγάλους ε, λιμένες και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δουλειά εκεί και μπορεί να δημιουργούν κάποιο επιπλέον άφθο ε, στα κάποια κράτη-μέλη και επηρεάζονται από αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε το θέμα. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω για το Ηνωμένο Βασίλειο, Στη σελίδα 42-43, τα τρία άτομα τα οποία ρωτήσατε για το Ηνωμένο Βασίλειο, εγώ εκπροσωπώ τη Σκοτία. Υπάρχει κάποια πτυχή που αφορά στη Σκοτία ή η φορέα συντονισμού είναι μόνο σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου. Μιλάτε για το τομεακό και εθνικό συντονισμό, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για τη σκοτική συνιστόσα, το οποίο δεν άκουσα εδώ. Ευχαριστώ πάντως για την έκθεσή σας και πάλι ζητώ συγγνώμη που δεν είναι εδώ όλοι όσοι από τους συναδέλφους θα ήθελα το θέμα είναι ότι είναι 6 παρά 20 το απόγευμα, ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει σε 9 το πρωί αυτή η παρουσίαση, μπορεί να ήταν ε, περισσότερη εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και περιμένω με ανυπομονησία τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλερ. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη μελέτη και θέλω να κάνω ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι πολύ σωστά η φάση δεν έχει περάσει, δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν κάνει λίγο πράγματα εδώ και θυμάμαι ότι η εποπτεία της αγοράς ήταν το βασικό βασικό θέμα σε μια προηγούμενη έκθεση στο οποίο επέμεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να έχω την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε αν πρόκειται να κινητοποιηθεί στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα τόσο καθυστερημένα. Ε, είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό το θέμα, τόσο ουσιαστικό για την Ευρώπη των πολιτών και των καταναλωτών και είναι κρίμα που δεν είναι περισσότεροι βουλευτές. Νομίζω ότι μπορούμε από κοινού να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που ανησυχούν τους ε, πολίτες μας. Εγώ επί δύο χρόνια ήμουνα υπουργό Γεωργίας και κατά τη Γαλλική Προεδρία ένα, υπέβαλα ένα μνημόνιο για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων που περνάνε τα εξωτερικά σύνορα. Παραδείγματο χάρη ε, προϊόντα από την Ουκρανία, ε, για, τα, για κάποια λάδια από την Ουκρανία κτλ. Υπάρχει όμως και το θέμα της ε, ισότιμης μεταχείρισης των παραγωγών. Η, και η ιδέα ότι στην αγορά μας δεν μπαίνουν προϊόντα που δεν σέβονται ε, ή σέβονται ελάχιστα ε, κανόνες που επιβάλλουμε στους δικούς μας παραγωγούς. Επομένως υπάρχει η ασφάλεια των καταναλωτών μας και η ισοτιμία μεταχείρισης για τους ε, παραγωγούς και τις θέσεις απασχόλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και είμαι ικανοποιημένος που το θέμα αυτό γίνεται προτεραιότητα της, του Μπαρόζου και της Σουηδικής Προεδρίας. Φυσικά το πακέτο αγαθών υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2008 και πολλά από τα μέλη αυτής της Επιτροπής, ε, η, η κυρία Σόλντε Μόζε και η κυρία Ανδρέας ε, που είναι εδώ, δούλεψαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια πιο, πιο ξεκάθαρη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Φυσικά δεν δούλεψαν μόνο αυτοί οι δύο συνάδελφοι, ε, δούλεψαν πολλοί βουλευτές Απλώς αυτή η Επιτροπή ε, έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον. Ε, και η κυρία Ρούλερ και άλλοι, θα μπορούσα να φέρω τους πάντες. Τώρα το θέμα είναι τι συνέχεια θα δοθεί σε όλη αυτή την προσπάθεια ε, και τι ερωτήσεις κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να μας πει, όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Ρούλερ, τι γίνεται, πώς δουλεύουν από κοινού αυτοί που είναι επιφορτισμένη με την ε, εποπτεία λιμένων και αερολιμένων. Μην ξεχνάμε τους αερολιμένες, ε, αυτούς που μπαίνουν ε, στα αεροδρομιά μας ε, και μην ξεχνάμε και αυτούς που μπαίνουν με χειραποσκευές, έτσι. Ε, πρέπει να θέσουμε ένα σοβαρό ερώτημα για να επαληθεύσει την ποιότητα της, του monitoring, τις καλές πρακτικές, την κοινή κατάρτιση των εθνικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τους έλεγχους αυτούς. Ε, αυτή η μελέτη ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα εν συνεχεία να μάθω αν η Κομισιόν θα μπορούσε να έρθει εδώ πέρα να λογοδοτήσει για ό,τι κάνει για, το, για την παρακολούθηση, το monitoring, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την κατάρτιση. ούτω ώστε οι διάφορες υπηρεσίες ελέγχου ε, να παίζουν το ρόλο τους ε, και να λειτουργούν τον ίδιο τρόπο. Κάτι άλλο ε, πολύ ενδιαφέρον η εξειδίκευση κάποιων προϊόντων για την εποπτεία κάποιων οικογενειών αγαθών. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε όλες οι χώρες να είναι επαΐουσες σε όλα τα προϊόντα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν κάποιες εξειδικεύσεις. Αυτές οι ιδέες που ήθελα να σας ε, υποβάλω και σας ευχαριστώ για την ποιότητα της έκθεσης ε, και της μελέτης. Ευχαριστώ. Κυρία Σαλντεμόζε, και συνεχεία θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Και εγώ ήρθα δυστυχώς καθυστερημένα στην παρουσίαση. Δεν ήξερα ότι είχαμε διεκπαιρεώσει τόσο γρήγορα τα προηγούμενα σημεία. Όπως είπε και η Κάθριν, τα περισσότερα κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν χωριστά κονδύλια για την εποπτεία της αγοράς. Το ερώτημα μου είναι, γιατί. Εσείς είπατε ίσως λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όταν δουλέψαμε επί του πακέτου αγαθών, είχαμε ξεκαθαρίσει ότι η εποπτεία της αγοράς είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί η εσωτερική αγορά σωστά. Χρειαζόμαστε περισσότερη εποπτεία από τα κράτη-μέλη της αγοράς. Επομένως, για να υλοποιήσουμε αυτά που είπαμε, νομίζω θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κονδύλια για την εποπτεία της αγοράς. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Δεν ήταν σαφή η νομοθεσία. Δεν ήταν καλή η νομοθεσία. Και μια επιπλέον ερώτηση. Τώρα που το πακέτο για τα αγαθά έχει εφαρμοστεί πλήρως, η εκτίμησή σας είναι ότι οι καταναλωτές θα είναι πιο ασφαλείς ε, στην Ευρώπη ή έχει παραμείνει απαράλλακτη η κατάσταση στην Ευρώπη. Και ένα ακόμα σχόλιο από τον κύριο Σβάμπ. Πολύ σύντομα θα απαραλλαχτη δηλαδή, η συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών ε, αρχών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς έχουν, έχει βελτιωθεί ή είναι αρνητικό το αποτέλεσμα. Η Κομισιόν. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν. Mr. McMillan. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε νόμιζα ότι η σύμβουλος ε, θα απαντούσε κάποιες ερωτήσεις πρώτα και μετά εγώ. Γι' αυτό αντέδρασα αργά. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι καλωσορίζουμε τη μελέτη και την έκθεση. Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε υποστήριξη προωθεί την εποπτεία της αγοράς, που είναι ένα θέμα που δεν ενδιαφέρει καθόλου για τους πολιτικούς. Νομίζω ότι θα έπρεπε να προωθηθεί ως θέμα προτεραιότητα στην Ευρώπη. Και κάποιοι από εμά εδώ θα θυμόμαστε πόσο σκληρά παλέψαμε να περάσει μέσα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, πρόσφατα μάλιστα. Οτιδήποτε λοιπόν δίνει υποστήριξη και ορατότητα στην ιδέα της εποπτείας αγοράς είναι ευπρόσδεκτο. Επίσης, από πλευράς Κομισιόν γνωρίζουμε ότι αυτή η μελέτη έγινε ε, με στενότητα χρόνου. Είναι κρίμα ίσως αυτό. Προφανώς ε, υπογραμμίζει σημαντικά θέματα, μέσα, πόρους, ε, ε, συγκεντρωτικές ή αποκεντρωτικές δομές, ο έλεγχος από τρίτες χώρες και η ανάγκη για καλές πληροφορίες. Από πλευράς μας στην Κομισιόν είμαστε κατά τη απογοητευμένοι. Και εδώ σας παραπέμπω σε μία από τις δύο ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές. Δηλαδή, ότι βρίσκουμε διάφορες δηλώσεις, το χάρη, ότι δεν υπάρχει χορήγηση πόρων, δεν θα δοθούν στο μέλλον πόροι, ας πούμε. Αυτός ο πίνακα σελίδα 19, Φερρυπίν, μου προκαλεί διάφορες σκέψεις και ερωτηματικά. γιατί είμαι πρόεδρος ε, της ομάδας εργασίας των κρατών μελών την ομάδα ανωτάτων υπαλλήλων, ε, εξειδικευμένων για την εποπτεία της αγοράς. Και περιέργως, εκεί μου δίνουν άλλα. Μάλιστα απαντήσεις, άλλα μου λένε εκεί. Ακούγονται πάρα πολλά για τις ανάγκες των κρατών μελών, ε, για τις σοβαρές ανάγκες και το γεγονός ότι δεν κάνουν κάποια πράγματα, δεν έχουν τους πόρους και τον προπολογισμό. Ε, συχνά λένε Εντάξει, η υποπτία της αγοράς σε εθνικό επίπεδο δεν είναι προτεραιότητα ούτω ώστε να πάρουμε κι εμείς ένα κομμάτι της πίτας του προϋπολογισμού. Φυσικά στους ε, consultants, στους συμβούλους λένε άλλα. Αλλά αυτά που μου λένε εμένα είναι η πλειοψηφία σε σχέση με αυτά που λένε σε εσά στον πίνακα 19. Άρα αυτοί που εφαρμόζουν το πακέτο αγαθών τι σχέση έχουν με αυτούς που λένε ε, τα όσα λένε στην, ε, στη μελέτη. Φυσικά δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρει κανείς απαντήσεις από εθνικούς εμπειρογνώμονες. Ε, ειδικά όταν φοβούνται ότι θα τους αφήσουν εκτεθειμένους εθνικές τους αρχές. Γιατί εθνικά δεν επιτρέπεται να λένε ότι δεν έχουν τα μέσα. Ίσως και αυτό είναι τμήμα της απάντησης. Αλλά τι, τι ξέρω εγώ. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια κάποια σύγχυση στο κείμενο της έκθεσης μεταξύ της ε, χρήσης ε, κάποιων εργαλείων, αξιολόγηση κινδύνου, ε, καθορισμό προτεραιοτήτων, το θέμα της δομής συγκεντρωτικής ή αποκεντρωμένης, τον έλεγχο των προϊόντων που μπαίνουν από τρίτες χώρες. Ο έλεγχος γίνεται πριν τεθούν στην αγορά ή μετά δεν είναι πολύ σαφή αυτά που γράφονται στην έκθεση, αλλά πιστεύω ότι η παρουσίαση που ακούσαμε πριν από λίγο είναι πιο σαφής. Για το θέμα του ράπεξ. Ότι πιστεύουμε ότι το σύστημα RAPEX υπάρχει και δεν είναι ίσως το πρόβλημα, το ράπεξ που έχει πρόβλημα, αλλά κάποιες εθνικές αρχές με τη χρησιμοποίησή του. Ίσως δεν έχουν τα μέσα να το χρησιμοποιήσουν. Ε, ίσως δεν έχουν την ίδια φιλοσοφία για το τι κοινοποιούν. Εγώ διάβασα στο κείμενό σα για κοινοποιημένα προϊόντα και τα μπερδεύεται με την ανείχνευση των επικίνδυνων προϊόντων. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω μπερδεύετε τα πράγματα λίγο στην έκθεσή σα. Οι συνάδελφοί μου ότι η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ μπορούν να πούν ίσω πολύ περισσότερα για το ράπεξ από ότι εγώ. Αλλά νομίζω ότι επικρίνουμε ένα εργαλείο το οποίο υπάρχει και είναι καλό. Ε, τόσο καλό που το βάλαμε και στον κανονισμό. Συλλογικά αποφασίσαμε, άρα να γνωρίζουμε ότι είναι καλό το εργαλείο. Ίσως λοιπόν δεν είναι τόσο λειτουργικό όσο θα έπρεπε αλλά ίσως αυτό να είναι θέμα ε, GPSD και όχι θέμα RAPEX. Οι συνάδελφοί μου στη ΣΑΝΚΟ ίσως μπορούν να συμπληρώσουν τα όσα είπα εγώ. Τώρα, η μεγαλύτερη απογοήτευσή μου είναι γύρω από τα μέσα. Αφορά τα μέσα. Ο στόχος ήταν να εντοπίσουμε τα βήματα που έλαβαν τα κρατη και αν ο στόχος της 1ης Ιανουαρίου υλοποιείται και αν έχουν και τα απαραίτητα, τους απαραίτητους σπόρους. Σα είπα ότι αυτό απόρα απέχει από τι πληροφορίε που παίρνουμε εμεί στην ομάδα εργασία από τα κράτη-μέλη. Ε, μπορώ να δεχθώ ότι λένε κάποια πράγματα στην ομάδα εργασία που δεν τα λένε δημοσία. Μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά νομίζω ότι το συνολικό μήνυμα τη έκθεση δεν τονίζει τα θέματα τα οποία είναι μείζωνα προβλήματα εφαρμογής. Εσείς εντοπίζετε κάποιες βέλτιστες πρακτικές ή καλέ πρακτικές, οι οποίες ενδεχομένως ε, δείχνουν ένα προσανατολισμό για μια μεταγενέστερη καλή συνεργασία, αλλά δεν μας λέτε τι λείπει. Και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο χρειαζόμαστε υποστήριξη. Ξέρουμε ότι πολλές εθνικές διοικήσει χρειάζονται υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι εξήγησε αυτό που ήθελα, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης σημειώνω διάφορα ερωτήματα ε, σε σχέση με τα μεγάλα λιμάνια. Είναι ένα σημείο το οποίο συζητάμε με τα κράτη-μέλη και ξέρουμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο τρόπο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, επιμερισμού των εθνικών πόρων μεταξύ των κρατών. Ε, δεν είναι μόνο θέμα ε, του Ρότερνταμ και του Αμβούργου. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα όταν 700.000 containers περνάνε ε, το χρόνο. Είναι τεράστιο νούμερο για να ελεγχθεί. Θα πρέπει κάπως να μοιράσουμε αυτό το βάρος στα κράτη-μέλη. Τις περισσότερες προσπάθειες των Ολλανδών, παραδείγματο χάρη, οι Ολλανδοί εστιάζονται εκεί, στους ελέγχους στα λιμάνια και όχι τόσο πολύ στην εσωτερική αγορά, γιατί εκεί έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ε, έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο από άλλα κράτη-μέλη. Αυτό το ξέρουμε. Επίσης ξέρουμε ότι εσείς μαζί με το Συμβούλιο βάλατε την ημερομηνία εφαρμογής 1η Ιανουαρίου του 2010 και θα θυμάστε ότι η Κομισιόν πίστευε ότι αυτή η ημερομηνία είναι ε, πολύ, πολύ σύντομη. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ήταν υπερβολικά αισιόδοξη αυτή η ημερομηνία και ότι η διαδικασία ε, εφαρμογής θα είναι πραγματική διαδικασία. Ε, τα κράτη-μέλη χρειάζονται χρόνο. Σε ορισμένα κράτη-μέλη πρέπει να γίνουν αναδιαρθρώσεις. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί συντονισμού. Τέλο πάντων, δεν θέλω να τα στυλιτεύσω τα κράτη-μέλη, να τα, να τα δακτυλοδείξω. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και δυστυχώ όλα αυτά δεν προκύπτουν από την έκθεση. Δεν βγαίνουν. Ξέρουμε ότι πολλέ προσπάθειε γίνονται Κάνουμε συναντήσεις ε, με τα κράτη-μέλη. Έχουμε και άλλη μία συνάντηση 15 Οκτωβρίου για να προσπαθήσουμε να οριστικοποιήσουμε το πώς τα κράτη-μέλη θα παρουσιάσουν τα εθνικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς. Ε, θα οριστικοποιηθούν ε, τον Οκτώβριο, ούτως ώστε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να έχουν έτσι τα προγράμματα και των άλλων έτοιμα για το 2010. Επίσης, το θέμα της αξιολόγησης κινδύνου και τα επικίνδυνα προϊόντα, για το αν υπάρχουν ε, διαφορές ε, ανάμεσα στον κανονισμό και στο GPSD, αυτά είναι τα θέματα δεύτερης προτεραιότητας. Προσπαθούμε να δώσουμε το σωστό προσανατολισμό προς το, προς το παρόν και μετά αυτά. Θα θέλαμε να δούμε τελικά, πραγματικά με ανυπομονησία, τι θα κάνετε με αυτή την έκθεση. Ελπίζαμε ότι θα μας υποστηρίξετε περισσότερο στο θέμα των μέσων και πόρων. Είμαι 100% πεπισμένος ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μακμίλαν από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Έχουμε επίσης από τη Γενική Διεύθυνση Σάγκο τον κύριο Σόρο ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να μας πει λίγα πράγματα για το RAPEX. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με όλα όσα είπε ο Ζακ Μακμίλαν. Πιο συγκεκριμένα μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ε, ότι η μελέτη αυτή φέρνει ένα τόσο αδιάφορο ζήτημα, όπως είπε και ο Μάρκ, ε, ενώπιον μιας πολιτικής συζήτησης. Ξέρουμε από καθημερινή πείρα ότι μπορεί να έχουμε εκπληκτικούς νέους κανόνες, αλλά οι κανόνες είναι καλοί αν υπάρχουν και οι πόροι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. όπως έλεγε και ο συνάδελφος, οτιδήποτε ε, δίνει προεπιξάρχοντα ρόλο στην εποπτεία της αγοράς, οποιαδήποτε πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να θέσουν ε, από τη θεωρία στην πράξη αυτά τα οποία διακηρύσουν, είναι πάντα χρήσιμο. όπως και οι θέσεις τις οποίες ε, λαμβάνει ο κλάδος ε, και η Όργαλιμ τώρα τελευταία που πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ε, συλλόγους βιομηχάνων και το ΆΝΕΚ που είναι η φωνή των καταναλωτών στην προτυποποίηση και την ασφάλεια των προϊόντων. Όλα αυτά είναι πρόσδεκτα και φυσικά θα ήταν και πάρα πολύ καλή ιδέα, δεν ξέρω αυτό το θέτω και σε εσά να οργανώσουμε κάποια στιγμή μια ακρόαση για την εποπτεία της αγοράς που θα περιλαμβάνει και την ProSafe η οποία είναι η κοινότητα για την, ε, των αρχών εφαρμογής ε, στα κράτη-μέλη και των καταναλωτών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Τώρα, για το RAPEX. Όπω έλεγε και ο Σάκ, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι, αλλά υπάρχει μια ουσιαστική παρανόηση για το ρόλο και τι λειτουργίε του συστήματο RAPEX ε, στη μελέτη. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί σαφεί ορισμοί στις κατευθυντήρε γραμμέ του RAPEX για το ποιο, είναι, ποιο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο προϊόν. Υπάρχουν ε, διεξοδικότατες κατευθυντήρες γραμμές για την αξιολόγηση κινδύνου, σοβαρή και πάρα πολύ σοβαρή κίνδυνη και ούτω καθεξής. Και φυσικά υπάρχουν και μία σειρά από λεπτομέρειες, ε, κάποιες από αυτές ε, ίσως και πιο σημαντικές, οι οποίες ε, επηρεάζουν κάπως το αποτέλεσμα της μελέτης. Είμαι βέβαιος ότι αυτό οφείλεται και στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έγινε η μελέτη, πολύ φιλόδοξο και είναι πολύ σημαντική η μελέτη για να ε, προαχθεί ο ρόλος της, ε, ε, της εποπτείας αγοράς. Ε, τα τρόφιμα, για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο του RAPEX ε, σε θέματα εποπτείας ε, της αγοράς. Το πλαίσιο για τα τρόφιμα, ευτυχώς, είναι πάρα πολύ διαφορετικό, πολύ πιο στεναρό από άλλα αγαθά. Σε καμία περίπτωση ε, δεν διακυβεύεται η ασφάλεια των προϊόντων ε, και πάντα θέλουμε να είναι αναλλαγική η αυστηρότητα. Ποτέ δεν θεωρούμε ότι ένα μπλουζάκι ή ότι μια ηλεκτρική συσκευή την χάνει της ίδιας αντιμετώπισης με το μοσχαρισιό κρέας. Αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ λέγοντας ότι Χαιρετίζουμε το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει αυτή η μελέτη προκειμένου να προβάλλει το ρόλο της εποπτείας της αγοράς. και να μας δώσει και κάποια, κάποιο μοχλό πίεση προς τις εθνικές κυβερνήσεις. Ευχαριστώ. Μήπως θέλετε να σχολιάσετε, κυρία Σίλβεστ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από την αρχή. Έγιναν αρκετά σχόλια. Ε, και ε, ξεκινώ με τον κύριο Κρόιτσμαν, ο οποίος δεν είναι πια εδώ, αλλά ο οποίος τόνισε τη σημασία των ε, ελέγχων στα λιμάνια. Δεν έχω να πω πολλά επ' αυτού, αλλά είναι ένα σημείο όπου θα πρέπει ίσως να αποδοθούν περισσότεροι πόροι στα λιμάνια δηλαδή και στα εξωτερικά σύνορα. Όντως, δίκιο έχεις αυτό. Και εσείς είχατε πολλές ερωτήσεις ε, τι σημαίνει ένα συντονιστικό όργανο ad hoc ε, κατά περίπτωση. Δεν σημαίνει ότι ε, πρόκειται για έναν οργανισμό αλλά για μια δυνατότητα συντονισμού όπου χρειάζεται. Δεν είναι δηλαδή ουσιαστικά ένα ε, συνηθισμένο όργανο. Επίσης είπατε γιατί τα κράτη-μέλη δεν αποδίδουν περισσότερους πόρους. Ουσιαστικά ε, οφείλονται δύο λόγοι τους οποίους μας ανέφεραν. Καταρχήν ότι ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη τουλάχιστον ευθύνεται η οικονομική κρίση και επίσης οι περισσότερες χώρες πιστεύουν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους με ανακατατάξεις πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν είναι αληθές αλλά αυτή είναι η γνώμη την οποία ακούμε από τις συνεντεύξεις. Μου ρωτήσατε ποια είναι η διάσταση. Δεν έχω πολλές λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά το Ηνωμένο Βασίλειο, αν κατάλαβα καλά, είναι πιο καλά οργανωμένο τομεακά και όχι, σε, ε, και όχι περιφερειακά. Οπότε χωρίς να μπορώ να το πω με βεβαιότητα υποθέτω ότι οι τομεακές αρχές επεμβαίνουν πιο πολύ. Μην το αναφέρετε όμως γιατί δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Η ερώτηση της κυρίας Ρούλε απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε θα την παρακάμψω. Η κυρία Σάλντερ Μόζερ έκανε ορισμένες ερωτήσεις ε, σχετικά με τους ε, πλεονάζοντες πόρους, ε, αλλά το κάλυψα. Επίσης είπατε εάν εφαρμοστεί η νομοθεσία θα είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω διότι υπάρχουν προφανώς προϋποθέσεις αλλά θα χρειαστούν και μεγάλη πόροι, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μας ελέγχθησαν. Άρα δεν είναι μια ερώτηση στην οποία μπορώ να σας απαντήσω. Ο κύριος Σβάμπ ρώτησε αν η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των ε, τελωνιακών αρχών έχουν, ε, έχει βελτιωθεί. Αλλά δεν έχουμε πολλά στοιχεία και φαίνεται δεν βλέπω δηλαδή μία έκθεση σχετικά με την ε, τάση που διαγράφεται. Θα ήθελα όμως να πω ότι σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχει πολύ συστηματικός συντονισμός μεταξύ των τελωνιακών αρχών και των αρχών εποπτείας αγοράς. Υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι μία συστηματική γενική αρχή. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε διερευνήσει επαρκώς και έτσι δεν μπορώ να σας αναφέρω λεπτομέρειες. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω σε ορισμένα θέματα τα οποία έθιξε ο κύριος Μακμίλαν. Δεν θα αναφερθώ στους πόρους, αλλά θα πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι αν κοιτάξουμε τον κατάλογο των συνεντεύξεων που έχουν επισυναυθεί στη μελέτη, νομίζω ότι ε, υπήρξαν 59 συνεντεύξεις και νομίζω ότι υπάρχει ένας αριθμός προσωπικότητων εκεί, οπότε ε, λυπάμαι εάν λένε άλλα πράγματα σε εμά και άλλα στην ομάδα εργασίας δεν μπορούμε να ελέγξουμε και μπορώ μόνο να βασιστώ στις ε, πεντενές συνεντεύσεις που κάναμε στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το ΒΑΠΕΞ, αν υπάρχουν παρανοήσεις, με συγχωρείτε, λυπάμαι. Αλλά ε, δεν ε, άκουσα ποιο ήταν το όνομα του εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, αλλά αντελήφθηκα ότι ε, ε, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις για, τις, ε, για τους δημόσιους διαγωνισμούς, για τις δημόσιες προμήθειες. Νομίζω όμως ότι με αυτά απάντησα σε ερωτήσεις σας και αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ακόμη εκρεμεί είμαι στη διάθεσή σας για να συμπληρώσω. Κύριε Μακμίλαν, έχετε σηκώσει, ζητά το λόγο, γι' αυτό σηκώσατε το στυλό σας. Με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε, αλλά ακούγοντας τις απαντήσεις αντελήφθηκα ότι εγώ δεν απάντησα σε δύο-τρία σημεία που έθιξαν ευρωβουλευτές, ε, δηλαδή ε, Καταρχήν δεν σας ε, καθιστούμε υπεύθυνους ε, για τις δηλώσεις των ε, επισήμων που άλλα λένε δημόσια και άλλα λένε ιδιωτικά. Ο κύριος όμως Μπαρνιέ αναφέρθηκε στην επιμόρφωση και στην εξειδίκευση σε ορισμένα κράτη, σε ορισμένους τομείς. Συζητείτε αυτό μεταξύ κρατών μελών για να συνδυάσουμε προγράμματα επ' αυτών των θεμάτων διότι γίνονται ήδη ορισμένες επιμορφώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των, ε, ε, προϊόν, των καταναλωτικών προϊόντων και μπορούμε να καλύψουμε όλο τον τομέα ε, του κανονισμού. Αλλά άλλο είναι αυτό το θέμα και άλλο να υπάρξει μια διαφορετική προτεραιότητα, δηλαδή για να υπάρξει η εφαρμογή, να ισχύσει το πρόγραμμα από πρώτη Ιανουαρίου με τις πρώτες προτεραιότητες απαιτεί και κάποια επιμόρφωση. Όσον αφορά την εξειδίκευση ορισμένων κρατών μελών, ακούσαμε πολλούς που ανέφεραν το θέμα αυτό και έχω ένα πρόβλημα. Η, η, ε, εθνικές κυβερνήσεις θα δεχθούν ένας επιθεωρητής από άλλο κράτος να επιθεωρήσει ε, στην επικράτειά τους ορισμένα προϊόντα που εισάγονται και αναφέρομαι εδώ στην γαλλική κυβέρνηση παραδείγματος χάρη θα δεχθούν οι ε, Γάλλοι εκπρόσωποι να επηρεάζουν τα γαλλικά αυτοκίνητα π.χ. εκτός Γαλλίας Δηλαδή ε, πώς μπορεί σε τεχνικό επίπεδο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς να υπάρξουν πολιτικές παρατυπίες διότι οι επιθεωρητές ε, της αγοράς προσπαθούν να εξετάσουν διάφορες ιδέες αλλά σαν ε, εθνικοί εκπρόσωποι τα δικά τους, οι δικές τους ευθύνες σταματούν στα σύνορα της χώρας η ιδέα λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Είναι μια ιδέα την οποία εξετάζουμε για να δούμε αν θα μπορέσουμε να την προωθήσουμε. Ο κύριος Σβάμπ είπε τι γίνεται με την ε, ε, συνεργασία μεταξύ τελωνίων και εποπτείας εσωτερικής αγοράς. Ε, για πολλές χώρες αυτό είναι ένα νέο θέμα και προσπαθούμε να πείσουμε τα κράτη ε, να ε, συνδέσουν ε, τους τελωνιακούς τους με τους υπευθύνους εποπτείας αγοράς αλλά μην ξεχνάμε ότι τα τελωνία είναι φορολογικές αρχές και θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία διότι μπορεί να μιλάμε για τον κανονισμό που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2000 και θα πρέπει οι τελωνιακοί να αντιληφθούν ότι είναι υπεύθυνοι και για την ασφάλεια. Χρειάζεται πολύ συντονισμός, αλλά υπάρχει κάποια κίνηση και όλα τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να κάνουν μία επιπρόσθετη προσπάθεια. Προσπαθούν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα επιτύχουν. Ευχαριστώ για τις επιπρόσθετες παρατηρήσεις σας. Για να καταλήξω, νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μια ακρόαση για την εποπτεία της αγοράς. Και εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτό το σήμα ασφάλειας ε, που ανέφερε ο κ. Σπαμπ και την πρόταση του κυρίου Μπαγνιέ, όπου το κάθε κρατός μέρος θα μπορούσε να εξειδικευθεί, ας πούμε, σε κάποιο τομέα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω ότι η νέα επιτροπή θα έχει αρκετή δουλίτσα.